So, dear Ας αρχίσουμε, λέει η πρόεδρος Κάμερ Εύερτ. Δεν έχει και πολύ νόημα να περιμένουμε περισσότερο. Ελπίζω ότι τα μέλη μας σιγά σιγά θα αρχίσουν να καταφθάνουν. Θα συνεχίσουν τα γερμανικά τώρα με την άδειά σας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσω στην ημερησία διάταξη θα ήθελα να απευθύνω το καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά σε ομάδα επισκεπτών την οποία έχει προσκαλέσει η συνάδελφός μας Julie Ward από την εκλογική της περιφέρεια και πρόκειται για μια οργάνωση που ασχολείται με τις τέχνες και λέγεται Jack Drum Arts. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να ε, σας ενδιαφέρει η σημερινή συνεδρίαση. Εκτός αυτού, με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω κοντά μας τον Επίτροπο κύριο Νάβρατσιτς. Γνωρίζετε ότι η σημερινή ανταλλαγή απόψεων αποτελεί μέρος του διαθρωμένου διαλόγου που διεξάγουμε ως Ευρωκοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, το 2017 τελειώνει σιγά σιγά καλά θα είναι να θα μπορέσουμε και να αναπαυθούμε λίγες ημέρες, αλλά πριν από αυτό είναι σωστό να γίνει μια καταγραφή ή μια απογραφή, αν θέλετε, των επιτευγμάτων των διαφόρων προγραμμάτων. Σημαντικό αυτό, διότι το 2018 θα αρχίσει η συζήτηση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την επόμενη γενεά προγραμμάτων. Είναι πολύ ευχαριστώ επίσης που πρόσφατα Έχουμε, έχει περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έγγραφο για την Ευρώπη του πολιτισμού και γνωρίζετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα λάβαμε και εμείς την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά και αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας η οποία ήδη κατ' επανάληψη έχει τονίσει τη σημασία της διάστασης αυτής και ήδη έχουμε καταθέσει και μελέτη για τις ευρωπαϊκές ταυτότητες, τις οποίες ε, με την ευρία είναι όχι ε, τα έγγραφα. Και μελέτη που είχαμε αναθέσει επίσης για τον εξυγχρονισμό της ανώτερης εκπαίδευσης. Θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση βέβαια και με την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν ώψη των ε, διαχωριστικών αυτών τάσεων και λαϊκιστικών τάσεων που διαπιστώνονται και εν ώψη της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη, είναι σημαντικό να τονιστεί ο κεντρικός ρόλος του πολιτισμού για μια γνήσια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και νομίζω ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτή είναι η εντύπωση που έχω αποκομίσει, αποτελεί ένα πρώτο και σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση όχι μόνο στη δική μας Επιτροπή και ούτε μόνο ε, στην ε, αρμόδια γενική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θεωρώ ότι όλοι στην Ευρώπη θα έπρεπε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με θέματα παιδείας, διότι η παιδεία θεωρώ ότι είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. Θα ακούσαμε πρώτα την ε, εισαγωγή σας και μετά θα έχουμε την ευκαιρία ελπίζω ότι θα έχω ε, μεγαλύτερη προσέλευση τότε, θα έχουμε την ευκαιρία να σας θέσω με ερωτήσεις, τις οποίες ε, θα ομαδοποιήσουμε αν δεν έχετε αντίρρηση και θα μπορείτε να απαντήσετε. Να σας δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο και, και να κάνετε την εισαγωγή σας. Thank you very much. Good morning. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω για να συζητήσουμε τις ε, προτεραιότητες σήμερα στον τομέα που μας απασχολεί. Η Ευρώπη ετοιμάζεται να πάρει μεγάλες αποφάσεις, θεμελιώδεις, για να καθορίσουν το μέλλον αυτής της Υπήρου και των λαών της. Τον υπόλοιπο χρόνο, μέχρι τις επόμενες ε, ε, εκλογές, πρέπει να αξιοποιηθούν. <clears throat> πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους για να αξιοποιήσουν τα δεδομένα της ζωής τους και να ενταχθούν σε ανθεκτικές οικονομίες και κοινωνίες. Θα πρέπει να διατηρήσει το χώρο της η Ευρώπη στον κόσμο. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν πήρε μια βασική θέση προς αυτό το στόχο. Εγκρίναμε ένα έγγραφο πολιτικής με φιλόδοξους στόχους συνεργασίας με τα κράτη-μέλη στην παιδεία και τον πολιτισμό. Χαίρομαι γιατί το όραμά μας εντάχθηκε στο, στις συζητήσεις των ηγετών στο, στη Σύνοδο Κορυφή στο Γκόθεμπορκ για τα κοινωνικά θέματα. Εμείς και αγραφούμε εκεί το όραμά μας για μια Ευρώπη που θα αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό της παιδείας και του ε, πολιτισμού χρησιμοποιώντας ανθεκτικές δομές ε, για ενεργό ταυτότητα και αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία. Θα δουλέψουμε προς μια Ευρώπη όπου η μάθηση, οι σπουδές, η έρευνα δεν θα μπλοκάρονται από διατάγματα. Ε, έτσι θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, καινοτομία και θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε θετικά τις κοινότητές μας. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει ευρωπαϊκή ταυτότητα, να την αισθάνεται ο πολίτης, ε, να νιώθει κομμάτι της κληρονομιάς μας. Οι στόχοι μας είναι δύσκολοι αλλά επιτεύξιμοι. Κάποια βασικά στοιχεία. Το όραμά μας ε, μιας, ενός γνήσιου χώρου παιδείας επικεντρώνεται στις ε, σπουδές και στους τίτλους σπουδών. Θέλουμε επίσης η κινητικότητα να γίνει πραγματικότητα για όλους τους σπουδαστές με υποστήριξη μιας φοιτητική ευρωπαϊκής κάρτας. Θα δουλέψουμε πάνω σε πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων βασικών, γλωσσικών, και ψηφιακών όπως και επιχειρηματικών δεξιοτήτων και να προωθήσουμε τη διαβίου μάθηση. Όλα αυτά χρειάζονται στέρεη χρηματοδότηση. Γι' αυτό η ανακοίνωση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο για να μπορεί να επιτύχει τους στόχους. Επίσης χρησιμοποίησαμε την ανακοίνωση για να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας να διαφυλάξουμε τις κοινέ αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά η οποία ε, ε, επεκτείνεται και στους δημιουργικούς τομείς. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ισχυρό ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τον πολιτισμό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευρωπαϊκή ποικιλομορφία και να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα που θα συμπληρώνει και θα εμπλουτίζει τις εθνικές και περιφερειακές ταυτότητες. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα, ελκυστικά και μας δίνουν εξαιρετική βάση για πρωτοβουλίες και δράσεις. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Πρόεδρο ε, της Επιτροπής για την πολύ θετική της αντίδραση στα σχέδιά μας. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και που έχω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ισχυρό σύμμαχο στην εφαρμογή της ε, ατζέντα η πρώτη ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτές τις φιλόδοξες ε, προσπάθειες είναι του χρόνου τον Ιανουάριο που θα γίνει η πρώτη σύνοδος κορφής για την εκπαίδευση. Θα συζητήσει θέματα χαμηλών επιδόσεων, κυρίως στις βασικές δεξιότητες. Η Σύνοδος Κορυφής θα συγκεντρώσει περίπου 400 συνέδρους, ε, τους καθήλυνα αρμόδιους υπουργούς και εμπλεκομένους όπως διδακτικό προσωπικό και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Είμαι πεπισμένος ότι η εκδήλωση αυτή θα είναι κλειδί για να ε, ενισχύσει περισσότερο την πολιτική συνένεση που χρειάζεται για φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. Ελπίζω ότι θα σταθείτε συμπαραστάτες μου σε, αυτό, σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Τώρα, ενημέρωση πιο λεπτομερή θα ε, σας δώσω, αρχίζοντας με την εκπαίδευση. Ε, το δύο σημαντικές ανακοινώσεις το Μάιο ε, αναφέρουν πώς μπορεί η Κομισιόν να, βοηθήσει τα κράτη-μέλη στον τομέα της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ε, σε ένα σεμινάριο ε, την επόμενη εβδομάδα θα αναπτύξουμε τα θέματα αυτά. Για τα σχολεία πιστεύουμε ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία στο επίπεδο των σχολείων. Έτσι τα σχολεία θα δίνουν υψηλή ποιότητα ε, σε ένα περιβάλλον ε, ένταξης, ενσωμάτωσης ε, και σε επίπεδο διδακτικού προσωπικού. Οι διευθυντές και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές θα είναι σε καλύτερη θέση. Το επάγγελμα θα θεωρείται έτσι πιο ελκυστικό. Ως παράδειγμα συγκεκριμένης δράσης που θα προλιάνει το έδαφος για μια πρωτοβουλία για την ψηφιακή μάθηση. Εμείς ε, στηρίζουμε τα σχολεία, ε, έχουμε ένα νέο selfie tool το οποίο ε, εισήχθη πιλωτικά σε 14 χώρες με μεγάλη επιτυχία. Το selfie δίνει ένα ενσταντανέ των σχολείων για το πού βρίσκονται και πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για τη βελτίωση του έργου τους. Το 2018 θα ξεκινήσει το εργαλείο. Στην εκπαίδευση θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις δεξιότητες και να προωθήσουμε την ανάπτυξή τους. Χαίρομαι διότι μια βασική δράση ήδη έχει αρχίσει. Αυτή τη βδομάδα οι Υπουργοί Εκπαίδευσης ε, έλαβαν απόφαση ε, για τους ε, αποφύτους που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν. Θα μπορέσουμε έτσι να συλλέξουμε στοιχεία και θα βοηθήσουμε τους σπουδαστές να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις και να, ε, θα βοηθήσουμε και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς. Τον επόμενο Ιανουάριο η Κομισιόν θα εγκρίνει μια σύσταση για να προωθήσει τις κοινέ αξίες για την εκπαίδευση και αναθεωρημένη ε, ε, παρουσίαση των βασικών δεξιοτήτων που χρειάζονται. Ένα άλλο θέμα είναι να προωθήσουμε τις κοινέ μας αξίες μέσα από την εκπαίδευση. Τα συστήματα εκπαίδευσης θα πρέπει να ε, μην έχουν αποκλεισμού. Θέλουμε να προωθήσουμε και μια ευρωπαϊκή διάσταση διδασκαλία. Να μάθουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι σπουδαστές και να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα. Δεν θέλουμε μια λύση και μια προσέγγιση ε, που θα εφαρμόζεται παντού για να διδάσκονται κάποια θέματα. Η εκπαίδευση όμως είναι ισχυρό εργαλείο που μπορεί να μας επιτρέψει να καταλάβουμε τα θεμέλια αυτής της πολιτικής κοινότητας της οποίας όλοι είμαστε μέλη. Η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμού είναι πολιτική προτεραιότητα για μένα. Πρέπει να φροντίσουμε κανεί να μην μείνει πίσω. Θα πρέπει να στηρίξουμε ιδιαίτερα ανθρώπους από μειονεκτικά περιβάλλοντα, με ειδικέ ανάγκες. Δυστυχώ ακόμα πόρο απέχουμε από το στόχο αυτό. Η τελευταία προσθήκη του Education and Training Monitor που δημοσιεύτηκε πριν από δύο εβδομάδες δείχνει ότι το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο είναι κυρίαρχο για να καθορίσει την ε, πορεία στις σπουδέ και στη ζωή των ε, νέων μας. Ε, στις 4 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσω τα αποτελέσματα του Monitor σε εσά για την νεολαία. Η μάθηση και η προετοιμασία για τη ζωή δεν γίνεται μόνο μέσα στη σχολική αίθουσα. Γίνεται μέσα από την εμπειρία, την αλληλεπίδραση, μέσα από άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση. Η Κομισιόν ετοιμάζει την αναθεώρηση μια στρατηγική για του νέου. Ε, το πλαίσιο για τη συνεργασία για την νεολαία. Θέλουμε να παρουσιάσουμε πριν από το επόμενο καλοκαίρι τι προτάσει μα. Η Κομισιόν θα στηρίξει τις προτάσεις στα στοιχεία που πήρε από τους ε, νέους ανθρώπους και τους εμπλεκόμενους με την νεολαία. Κάνουμε αξιολόγηση της τωρινής μας στρατηγικής για να προβληματιστούμε για το μέλλον. Χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνει ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και προσβλέπω στην ε, έκθεση της ε, κυρία Σέινταρ για τις προτάσεις για το μέλλον. Ε, η προτεραιότητά μου για την πολιτική για τους νέους είναι να δημιουργήσω με ευκαιρίες τους νέους να ενταχθούν, να εμπλακούν, να μεγαλώσουν ως ανθρώπινα όντα, να στηρίζουν τους άλλους. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη αυτού του στόχου. Από τότε που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, πάνω από 41.000 νέοι άνθρωποι εγγράφηκαν για το σώμα, δείχνοντας ενθουσιασμό και αλληλεγγύη όπως και βούληση να βοηθήσουν ανθρώπους σε ανάγκη. Αυτό με κάνει πολύ περήφανο. Τη Δευτέρα οι Υπουργοί Νεότητας ε, συμφώνησαν με την πρότασή μας για μια νέα νομική βάση για το σώμα αλληλεγγύης. Χαίρομαι που κάνατε ό,τι ε, ε, ε, χαίρομαι διότι το Κοινοβούλιο έλαβε θέση για να αρχίσει ο τριμερής διάλογος γρήγορα. Θέλουμε να φτάσουμε γρήγορα σε πολιτικές αποφάσεις ώστε η νομική βάση να εγκριθεί το ταχύτερο δυνατόν το 2018. Εμεί θέλουμε για χάρη των νέων να κινηθούμε γρήγορα. Πάμε στον πολιτισμό τώρα. Θα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες θα εγκαινιαστεί το έτος ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ και εδώ για την υποστήριξη. Για το... Ε, έχω μεγάλες φιλοδοξίες για το έτος. Θέλω η πολιτιστική κληρονομιά να επιβεβαιωθεί ως εγκάρσια πολιτική και θεμελιώδες κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, επικεντρωνόμενος σε τέσσερις αρχές ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Εμπλοκή, βιωσιμότητα, καινοτομία και παραγωγή. Πολλά έχουν γίνει ήδη για να προετοιμαστούμε για το ευρωπαϊκό αυτό έτος. Αρχίσαμε ε, ειδική ε, πρόσκληση για προγράμματα συνεργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και πήραμε πολλές αιτήσει, ε, εντυπωσιακό αριθμό. Πετύχαμε να κινητοποιήσουμε τους εμπλεκόμενους στην πολιτιστική κληρονομιά σε όλη την Ευρώπη και να τους συνδέσουμε με τους εθνικούς συντονιστές για αυτό το θέμα. Συνδεθήκαμε και με νεολαίστικες οργανώσεις ε, το έτος αυτό είναι μια πρωτοβουλία από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση. Θέλουμε να έχουμε επαφή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με τον κόσμο. Σε ενωσιακό επίπεδο κινητοποιούμε διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν για συνεργασία. Συνεργασίες που θα συμπεριλάβουν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, πολλές εκδηλώσεις, ε, διακρατικά προγράμματα και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες υψηλής ορατότητας πολλά πρέπει να γίνουν για να, έχουμε, ε, να, να αφήσει μια κληρονομιά το έτος αυτό. Θα δουλέψουμε με όλες τις οργανώσεις εταίρους και κράτη-μέλη και θεσμικά όργανα της Ένωσης. Το έτος αυτό είναι πραγματικά γνήσια ευρωπαϊκό έργο. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκή ταυτότητα και καλύτερο μέλλον. Ε, τώρα, πέρα από τα σύνορά μας, παράλληλα με τη στρατηγική για τις ε, διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, δουλεύουμε για να ε, αναδείξουμε στις εξωτερικές σχέσεις τη διάσταση του πολιτισμού, ενθαρρύνοντας πολιτιστικές σχέσεις με τις χώρες εταίρους και προκρίνοντας τις άμεσες επαφές μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο γιατί ήταν από τους ισχυρότερους υπέρμαχους μιας πολιτιστικής πολιτικής εξωτερικών, πέραν των συνόρων. Ε, δουλεύουμε προς ε, μια σταδιακή στρατηγική προσέγγιση για να ενισχύσουμε τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Είμαι σίγουρος ότι μέσα σε ένα χρόνο θα έχουμε μια ε, κοινή στρατηγική που θα συνενώνει πόρους και θα έχει πολλαπλασιαστικό όφελος. Σχετικά τώρα με τις πολιτιστικές δημιουργικές τέχνες και βιομηχανίες, από το 2006 υπάρχει πολιτική η οποία ε, βάζει την αξία της δημιουργίας στο προσκήνιο και ε, δημιουργεί ε, κονδύλια για χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά χρηματοδοτικά μέσα στο, για το μέλλον πρέπει να συνεργαστούμε ώστε η υποστήριξη στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα θα τους επιτρέψει να αναπτυχθούν συμπεριλαμβάνοντας εκείνους τους τομείς που είναι πιο ευάλωτοι και εξαρτώνται πολύ από την ε, δημόσια ε, χρηματοδότηση. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στον τομέα της μουσικής. Περισσότερο από τους άλλους δημιουργικούς κλάδους, αυτός ο τομέας ε, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα λόγω της ψηφιοποίησης. Αυτό οδήγησε σε καινούρια επιχειρηματικά μοντέλα, αλλαγή παραγωγής στην κατανομή, στη διανομή, στην κατανάλωση Εμεί κάνουμε εντατικό διάλογο με τον τομέα και είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να αναπτύξουμε σε συγκεκριμένη προσέγγιση στη μουσική, ε, οικοδομώντα πάνω στα βασικά στοιχεία δημιουργικότητα, ποικιλομορφία, ανταγωνιστικότητα. Τα έχει αυτά ο κλάδο. Υπ' αυτή την έννοια χαιρετίζω το έργο τη Επιτροπή που μα βοήθησε να στηρίξουμε καλύτερα και να προωθήσουμε τον τομέα τη μουσική. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τι προτάσει τη Κομισιόν για προπαρασκευαστική δράση. Ε, ε που προάγει ταλέντα και την ποικιλομορφία στη μουσική. Αυτό είναι σημαντικό για να τεστάρουμε νέες προσεγγίσεις και ε, αυτό θα το κάνουμε σε αρχές του 2018 η δράση που προγραμματίζομαι θα μας βοηθήσει να προβληματιστούμε και να καταλήξουμε σε πιο στοχευμένη υποστήριξη της μουσικής στο νέο πρόγραμμα μετά το 2020. Ε, υπολογίζομαι στη συνεχιζόμενη υποστήριξη αυτής της Επιτροπής για την πρωτοβουλία της Κομισιόν για τη Μουσική. Αθλητισμός τέλος. Ο αθλητισμός φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Αυτό φάνηκε και από τη βδομάδα αθλητισμού από τις 23 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό αποδείχθηκε εκεί. Ε, πριν από τρία χρόνια είχε γίνει κάτι παρόμοιο. Είναι πάρα πολύ ε, ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι η ιδέα αυτή έχει προχωρήσει και έχει εγκριθεί πολύ γρήγορα και υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη. Φέτος μαζί με τους ε, συναδέλφους Αντριουκάητη και Χόγκαν ξεκίνησα μια νέα πρωτοβουλία. Θα δουλέψουμε οριζόντια, διατομεακά για να προωθήσουμε υγιεινό τρόπο ζωής ο αθλητισμός έχει μεγάλη δύναμη στις κοινότητες. Ε, εδώ παίζουν ρόλο και τα αθλητικά βραβεία που αναγνωρίζουν τις οργανώσεις που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό για να μειώσουν τις, ε, την περιθωριοποίηση ε, μειονεκτικών ομάδων. Θα γίνει, πέρσι έγινε η απονομή των βραβείων. Τέλος, δύο λόγια για τις εκστρατείες για την 30η επέτειο του Εράσμους. Αυτή η επέτειος μας ε, επέτρεψε να δώσουμε την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία, τον αθλητισμό μέσα από το Erasmus Plus. Δείξαμε τον επιτυχή ρόλο που παίζει αυτό το πρόγραμμα για να αντιμετωπίσει τις ε, πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη πάνω από 900 εκδηλώσεις και τεράστια συμμετοχή των κοινωνικών μέσων και του τύπου. Η εκστρατεία αυτή έφτασε σε πάνω από 90 εκατομμύρια Ευρωπαίους μέχρι τώρα. Ε, πολλοί πέρα από αυτούς που ωφελούνται από το πρόγραμμα. Ε, το κλείσιμο ή τη, ε, τελετή, η τελετή κλεισίματος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Με αυτή την ευκαιρία θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τον ενθουσιασμό με τον οποίο υποστηρίξατε σε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις της Κόση Κομισιόν. Φέτος είναι θαυμάσια ευκαιρία να, έχουμε, να αναπτύξουμε κοινό όραμα για το μέλλον του προγράμματος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βελανσφέρ και τους σκιώδες που συμμετείχαν στην, στην έκθεση υλοποίηση του Erasmus Plus και όλους εσάς που συμμετείχατε στο Στρασβούργο στον Ιούνιο σχετικές εκδηλώσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την πολύτιμη συμβολή σας και στην, ε, στην, στην ε, Ολομέλεια ε, που επέτρεψε το Erasmus Plus να υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο. Είστε καθοριστικοί στο να βοηθήσετε να χαράξουμε το μέλλον σε αυτούς τους τομείς στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, πραγματικά ε, πολύ εκτεταμένη η επισκόπηση που μας δώσατε για τα πολλά θέματα του χαρτοφυλακίου σας. Ως συνήθως θα δώσω τον λόγο στους συντονιστές και συντονίστρες για τρία λεπτά. Μετά θα απαντήσει ο Επίτροπος και μετά θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο και άλλα μέλη που έχουν ήδη ζητήσει να λάβουν το λόγο και πρώτα η κυρία Σαμπίνε Φερχάιεν. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μας διαθέτεται χρόνο για διάλογο σήμερα. Νομίζω η ανακοίνωση που εκδώσατε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια σωστή αφετηρία ιδίως δηλαδή η προσπάθεια ενίσχυσης ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της παιδείας. Σημαντικό θέμα, το οποίο ε, επεξεργαζόμαστε εμείς εντατικά εδώ και πολλά χρόνια για να αξιολογήσουμε διάφορες μεθόδους για την τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Και από τα πιο σημαντικά προγράμματα προς το σκοπό αυτό είναι το έρασμο ΣΥΝ. Και ξαναλέμε ότι είναι ένα θαυμάσιο πρόγραμμα το οποίο δυστυχώς υποχρηματοδοτείται. Ερώτηση λοιπόν για το μεσοπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σημαντική αύξηση του προπολογισμού του Ερασμοσύν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Το ίδιο ισχύει για το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Επίσης υποχρηματοδοτείται σημαντικά προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να προωθηθούν και δεν χρηματοδοτούνται παρκώς. Θα προωθήσει τις απαιτήσει αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στο Συμβούλιο Υπουργών. Άλλο θέμα είναι η ψηφιοποίηση. Ειδικώ για την παιδεία, σε πολλούς τομεί βλέπουμε να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις δεξιοτήτων και προσόντων. Η νέα γενεά γνωρίζει να χειρίζεται τα μηχανήματα, αλλά τι γίνεται με την ικανότητα αναζήτησης νέων ειδήσεων, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή χρειάζεται υποστήριξη και εκπαίδευση και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών. Πρέπει όμως να δοθούν κατευθύνσεις και υποστήριξη για τους τομείς εκείνους που και εμείς κρίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικοί. Άλλο σημαντικό θέμα είναι για μένα το κατά πόσον για την προώθηση των creative industries θα μπορέσουν να δοθούν ενισχύσεις όχι μόνο στα προγράμματα πολιτισμού κλπ αλλά και μέσω των διαφρωτικών ταμείων με πιστώσεις που διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιες πιστώσεις να διατεθούν και σε αυτούς που δημιουργούν πολιτιστικό περιεχόμενο. Από τη δική μου περιφέρεια γνωρίζω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να χρηματοδοτηθεί κανείς ως καλλιτέχνης από πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ακόμα και αν έχουν ε, συνεταιριστεί οι καλλιτέχνες αυτοί. Πώς είναι δυνατόν σε συνεργασία με άλλους επιτρόπους να φτιάξετε ένα είδος master plan, ένα βασικό σχέδιο δηλαδή, το οποίο να επιτρέψει να ανοίξουν οι χρηματοδοτήσεις και γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ τον Επιτροπό για την ανακοίνωση εν ώψη της διάσκεψης κορυφής θα ήταν παράξενο ή παράδοξο να μην δείξουν η Κομισιόν ή το Συμβούλιο ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι ένα αποσπαστό τμήμα της κοινωνική διάστασης της Ευρώπης. Όταν είχαμε δει το θεματολόγιο δεν υπήρχε και χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που το Συμβούλιο και η Κομισιόν παρουσίασαν προτάσεις. Αυτό όμως αφορά και αυτό που λέγατε πριν εσείς προηγουμένως, ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η Κομισιόν στο σύνολό της θα αλλάξει βηματισμό και την ανακοίνωση τη συμμεριζόμαστε βεβαίως, παρόλο που δίδεται λιγότερη προσοχή στο πολιτιστικό τμήμα, αλλά τέλος πάντων το καλύψατε αυτό σήμερα στην ομιλία σας. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Κομισιόν που δεν έχει τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στις 10 προτεραιότητες της, χαίρομαι που ακολουθεί αυτή την προσέγγιση τώρα. Αυτό που θέλαμε δηλαδή εμείς και χρόνια. Θα αφήσω τη συναφόρη Βάσκα να εμβαθύνει για τα θέματα εκπαίδευσης και να πω τα εξή. Χαιρόμαστε που επιτέλου θα υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης, όπως είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να αναθεώσουμε κάποια συστήματα, θα πρέπει να προωθήσουμε την κινητικότητα των μαθητών και των φοιτητών και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και στα πλαίσια της εφαρμογής του θεματολογίου για τις δεξιότητες που στην ουσία αποτελούν κομμάτι αυτής της τέταρτης τεχνολογικής επανάστασης που ζούμε. Είδα στην ανακοίνωσή σας γίνεται λόγος για μια συνεργατική παρέμβαση σε συνεργασία δηλαδή με την Γενική Διεύθυνση Connect στα πλαίσια του Digital for Culture όπως είχε ανακοινωθεί. Επίσης υπάρχει και το θέμα το να δοθούν ευκαιρία στους διδάσκοντες και στους νέους επαγγελματίες ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες που υπάρχουν. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία που θα πρέπει να υποστηρίξει η Κομισιόν με το e-learning, το e-teaching, όλα αυτά τα εξαποστάσεως μορφές δασκαλίας και μάθησης. Εμείς ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο την ενίσχυση των κονδυλίων του Εράσμους. Θα θέλαμε να υπερδιπλασιαστούν. Και στο πρόγραμμα του κυρίου Γιούνκερ γίνεται λόγος για να φτάσουμε στο 30% των νέων που θα συμμετέχουν στο Εράσμους μέσω και ιδιών πόρων και υπάρχει και μια μάχη αυτή τη στιγμή και μια ισχυρή δέσμευση εκ μέρου τη Γενική Διεύθυνση ώστε αυτό να υλοποιηθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή καλύπτουμε μόνο το 4% των νέων. Τώρα για το θέμα που αναφέρατε, για του πολίτε, του εθελοντέ. Ένα λεπτάκι να το τελειώνω, ναι. Έχουμε μια μεγάλη ανησυχία που αφορά κάτι το ενδιαφέρον αλλά και την αλληλεγγύη. Εσείς είπατε ότι θέλετε σύντομα να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Όμως με ανησυχεί αυτό γιατί την τελευταία φορά η πλειοψηφία του Συμβουλίου δεν αποδέχτηκε την ιδέα του 25% νέων πόρων, δεν αποδέχτηκε το να πάρουμε πόρους από άλλα προγράμματα και να μείνουμε μόνο στο Erasmus. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια νέα συμφωνία και επιμένουμε προς αυτήν την κατεύθυνση εμείς Κοινοβούλιο. Και κλείνω η δημιουργική Ευρώπη και εκεί υπάρχουν πολύ λίγοι πόροι και κατακαιρματισμός διαχείρισης. Ευχαριστώ. Η Ευχαριστώ. Η κυρία Χιμένεθ ναι. Να μιλήσω για την επιστήμη ως πολιτιστική κληρονομιά όλων των Ευρωπαίων και ως πυλώνα δημιουργίας αυτού του, αυτού του είδους ε, σχέσεων και δεσμών στην ευρωπαϊκή ταυτότητα. Παλιά ούτε καν δρόμους είχαμε, που να είχαμε και ίντερνετ μάλιστα. Πάντως υπήρχε όμως μια ισχυρή επαφή μεταξύ των διαφόρων επιστημόνων που αντάλλασαν αποτελέσματα ερευνών ή απόψεις και θεωρείται ότι Σήμερα αρκούν όλα αυτά ώστε ο Ευρωπαίος πολίτης να θεωρήσει την επιστήμη ως τμήμα της ε, πολιτιστικής του κληρονομιάς και να απολαύσει αυτή. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ο κύριος Σόλτης. Ο κύριος Χουντής, να με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Ομολογώ ότι είχατε μια δύσκολη προσπάθεια, διότι κατά την άποψή μου έχετε να διαχειριστείτε αμφιλεγόμενες έννοιες και ιδέες και πολιτικές θα έλεγα. Κύριε Επίτροπε, όπως γνωρίζετε στην αρχαία Ελλάδα από τα βασικά μαθήματα εκτός από τη ρητορική ήταν και η διαλεκτική. Παρεπιπτόντως ήταν και η μουσική και χάρηκα που υπάρχουν αναφορές στη μουσική αλλά δεν έχω τον χρόνο να αναλύσω τι προβλήματα και τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό αν θέλουμε να προσεγγίσουμε ορισμένα ζητήματα. Η διαλεκτική λοιπόν λέει διάλογος. Ο χρόνος δεν με επιτρέπει να σας πω την άποψή μου σε αυτά που αναλύσατε. Επομένως υπό τη μορφή ερωτήσεων να σας ε, θέσω πώς θα αντιλαμβάνομαι αυτά. Πρώτο ερώτημα. Μιλάτε, το έχω διαβάσει το κείμενο και η ανάλυση σας ήταν ε, καλή ως προς αυτό. Μιλάτε για την συμβολή της εκπαίδευσης, για την αναζήτηση ή ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ερώτηση πρώτη. Ποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα, κύριε Επίτροπε. Είναι αυτή που αναζητούμε στις συνθήκες ή είναι τα διλήμματα που έχουμε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αξίες όπως ανταγωνισμός ή αλληλεγγύη, δημοκρατία ή μονόδρομος, κοινωνικά δικαιώματα ή δημοσιονομική πειθαρχία. Σας παρακαλώ, δώστε μια απάντηση. Τα κείμενα είναι γενικόλογα. Η χρήση αυτού, δωστε μια απαντηση τα κειμενα ειναι γενικολογα η χρηση αυτου του ζητήματος είναι ad hoc. Δεύτερη ερώτηση. Σε κάποιο σημείο αναφέρατε ότι υπάρχουν, ε, αν το συγκράτησα καλά, διατάγματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της παιδείας, της έρευνας. Μπορείτε να μου πείτε τι εννοείτε ως προς αυτό. Σπέβδω να σας δώσω μια δική μου εκτίμηση. Ότι αυτό που εμποδίζει την πραγματική παιδεία, την εκπαίδευση, είναι οι πολιτικές της λιτότητας, η υποχρηματοδότηση της δημόσιας παιδείας, η υποχρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως φάνηκε από την συζήτηση που έχουμε κάνει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην έχουμε και τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς. Δεν θέλω να σας αναφέρω στοιχεία από την Ελλάδα γιατί δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό αναρωτιέμαι, η Γαλλία από όσο ξέρω έχει μεγάλο πρόβλημα με το εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν μπορεί να πάρει εκπαιδευτικούς διότι πρέπει να είναι εντάξει με το έλλειμμά της. Επομένως αυτό που εμποδίζει την ανάπτυξη κατά τη γνώμη μου είναι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές και οι πολιτικές των περικοπών κοινωνικών ταπανών και υποχρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων. Και τρίτη ερώτηση για να μην σα κουράζω. Αναφερθήκατε σε κοινέ αξίες για την παιδεία και σε κάποιο σημείο πάλι το αμφιλεγόμενο θέμα περί αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Ερώτηση κύριε, ε, κύριε Επίτροπε. Μέσα στις δεξιότητες ή μέσα στην αξιολόγηση το τι μαθαίνουν τα παιδιά, οι φοιτητέ, αναφέρεται και η επιδόση τους στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδέ. Αναφέρονται τα ζητήματα των αξιών, αναφέρονται τέτοιες επιδόσεις ή είναι οι τεχνικές επιδόσεις που απαιτεί η αγορά προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματική, άρα να έχει περισσότερα κέρδη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για, Για τα ψηφιακά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις παλαιές μεθόδους. αρχίσαν ήδη από το δημοτικό στην Γαλλία, αρχίσαν να καταργούν ακόμα και τον πολλαπλασιασμό και την προπαίδεια και μετά διαπίστωσαμε ότι δεν απέδιδε η προσπάθεια αυτή. Και οι νέοι τώρα που γράφουν SMS και όλα αυτά με το διαδίκτυο γράφουν συνεχώς ανορθόγραφα. Καταργούν τις λέξεις, γράφουν τις μισές ενώ τα παιδιά έχουν στο σπίτι τους το απαραίτητο υλικό, νομίζω οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει να τους μάθουν ξανά τα θεμελιώδη. Βεβαίως η έρευνα διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου για να κάνουν έρευνα τα παιδιά δηλαδή. Τώρα για την ταυτότητα του σπουδαστή, την ευρωπαϊκή ταυτότητα του σπουδαστή, έχω μια ερώτηση. Αυτό επιτρέπει να λαμβάνουν χρήματα, επιτρέπει να πάνε σε πανεπιστήμιο. Δεν έχω καταλάβει καλά. Και τέλο για την διεθνή κατάταξη των πανεπιστημίων. Λέτε ότι μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα η Ευρώπη. Εμεί προσπαθήσαμε στη Γαλλία να συνενώσουμε τι μεγάλε σχολέ να ανταλλάξουν απόψει και να συνεργαστούν. Μέχρι τώρα όμω δεν έχει αποδώσει η προσπάθεια αυτή, διότι κάθε μεγάλη σχολή, πανεπιστημιακή δηλαδή, θέλει να τηρήσει, να κρατήσει δηλαδή τη δική της και ε, τη δική της ταυτότητα και δεν θέλει να αναμειχθεί με άλλες. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Πριν επιστρέψω το μικρόφωνο στον κύριο Επίτροπο για να απαντήσει, θα ήθελα να προσθέσω μια ερώτηση. Ήλπιζα να την κάνει κάποιος άλλος βουλευτής, αλλά θα την κάνω εγώ. Διαβάζοντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα σχετικά ε, δελτία, fact sheet, ξεπηδούν ορισμένα ερωτήματα για το πρόγραμμα για το μέλλον της Ευρώπης μου φαίνεται σαν να πρόκειται για νέο πρόγραμμα ευρωπαϊκό προώθησης των πολιτιστικών και της δημιουργικής βιομηχανίας και ένα πρόγραμμα συνέχειας για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση σκέπτεται να χωρίσει δηλαδή το Creative Viewer πρόγραμμα ένα οπτικοακουστικό και ένα πολιτιστικό τμήμα. Εσείς μιλήσατε και η αύξηση των κονδυλίων στο πρόγραμμα Έρασμος. Αλλά δεν λέτε τίποτα για το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Και ενδεχομένως για τα δύο υποπρογράμματα, εάν χωριστεί. Μπορείτε να πείτε λίγα λόγια σχετικά. Προς ποια κατεύθυνση δηλαδή κινείται ο προβληματισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Ναύρατσιτς Προσπαθήστε να δω, θα τα καταφέρετε, να απαντήσετε στις πολλές αυτές ερωτήσει ερωτήσεις μέσα σε πέντε λεπτά. Ξέρω ότι θα είναι δύσκολο. Θα τηρήσω την πειθαρχία ώστε να μείνει χρόνος και για τον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ακόμα συντάσσουμε το σχέδιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καμιά φορά λοιπόν μετακινούνται οι θέσεις. Διαμορφώνεται μια γενική συνένεση πάντως για περισσότερη χρηματοδοτική υποστήριξη για το έρασμο ΣΥΝ. Αυτό φάνηκε και στην κοινωνική διάσκεψη κορυφής του Γκότενμπουργκ μεταξύ των χώρων μελών και μου φαίνεται σημαντικό βασίζομαι και στην υποστήριξή σας. Είσαστε φυσικός μου σύμμαχος για να κάνουμε τον αγώνα για περισσότερα χρήματα για το έρασμο Θα θέλαμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του έρασμο ΣΥΝ ώστε να καλύψει και άλλες κοινωνικές ομάδες λιγότερο προνομιούχες όσον αφορά το οικονομικό του υπόβαθρο. Να φτάσουμε δηλαδή στην κοινωνική διαστρωμάτωση και στους ανθρώπους εκείνους που δεν είναι της ανώτερης μεσαίας τάξης αλλά και της ε, μεσαίας και της χαμηλότερης μεσαίας τάξης ας το πω έτσι και ακόμα πιο κάτω να φτάσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα πρόσωπα γιατί είναι σημαντικό εργαλείο για την κοινωνική συμπερίληψη. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον συν λοιπόν περισσότερο για να ενδυναμώσουμε τους νέους ανθρώπους που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχες οικογένειες. Έχει κάνει μια παρατήρηση η κυρία Φερχάιν χωρίς μικρόφωνο όμως. Το πρόγραμμα Comenius δηλαδή για να ενισχύσουμε την κινητικότητα <clears throat> μαζί με την ηλεκτρονική ή e-training, που είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μιλώ για ε, μαθητές της ε, δευτερεύουσας της, ε, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τα ψηφιακά συζητούμε πολύ πώς να υποστηρίξουμε τις χώρες μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστέ στην κριτική σκέψη. Γιατί η κριτική σκέψη είναι και το καλύτερο όπλο απέναντι στις ψευδείς ειδήσει και να μπει στα εθνικά προγραμμάτα διδασκαλίας για να μπει και στην τυπική και στην άτυπη και στην μη τυπική εκπαίδευση αναπτύσσοντας policy instruments, οργανώνοντας εργαστήρια, προωθώντα τι καλύτερε πρακτικέ μεταξύ των χωρών μελών. Προσπαθούμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τις ψευδείς ειδήσει αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη. Η δημιουργική ε, βιομηχανία, αυτό το creative industry, είναι πολύ σημαντική υπόθεση και συνδυάζεται και με τη μεταρρύθμιση του copyright και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να ενισχύσουμε την creative industry για να δημιουργήσουν δηλαδή οικονομικό, ε, να δημιουργήσουν, να δημιουργήσουν πολιτιστικό περιεχόμενο. Εκδώσαμε εκθεσή στην οποία περιλάβαμε και τις δράσεις και τις συνθήκες πλαίσια για την ενίσχυση της καινοτομίας την πρόσβαση της creative industry σε χρηματοδοτήσεις, θέσπιση βραβείων και το πρόγραμμα για την στήριξη του, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βάζουμε τα θεμέλια δηλαδή τώρα για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την δημιουργική βιομηχανία. Βρισκόμαστε όμως σε ένα σημείο τομής της βιομηχανικής πολιτικής και της πολιτιστικής πολιτικής. Και καμιά φορά ανταγωνίζονται μεταξύ τους οι τομείς αυτοί. Και είναι δύσκολο να προωθήσουμε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για την βιομηχανία δημιουργή, ε, καλλιτεχνικής δημιουργίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμφώνησε το Συμβούλιο σε μια συνολική αντίληψη. Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός. Προχωρούμε στον τριμερή διάλογο και πιστεύω ότι, γιατί υπάρχουν πολλοί, πολλά ευαίσθητα θέματα εκεί, πολλά ευαίσθητα θέματα τα οποία θίγει μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και το Συμβούλιο, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής. Είμαστε ανοιχτοί όμως για να κάνουμε συμβιβασμούς και να σας υποστηρίξουμε και εσάς να μπορέσετε να εξεύρετε συμβαστικές λύσεις με το Συμβούλιο. Του χρόνου θα είναι το έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για μας και θέλω να ε, ρίξουμε το φως σε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες, στις τοπικές κοινότητες. Δεν γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. Ακόμα Τώρα, ένας Ισπανός δεν γνωρίζει τα βασικά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς των Βουλγάρων, για παράδειγμα. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό στοιχείο της παράδοσης που εν τέλει δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα τμήματα της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς. Και καλούμαστε να ανακαλύψουμε αυτή την κληρονομιά, να αναδείξουμε τα στοιχεία αυτά της πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαφόρων κοινοτήτων. Θα βασίσω λοιπόν τις εκδηλώσεις του επομένου έτους στο τοπικό επίπεδο και ελπίζω ότι θα προσφερθούν έτσι σημαντικές ευκαιρίες στις τοπικές κοινότητες να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα προβολής για την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το κείμενό μα για την ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι λόγο, διότι νομίζω ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο. Υπάρχουν διάφορα στρώματα ταυτοτήτων. Τοπική ταυτότητα που είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη. Περιφερειακή ταυτότητα, κάπω λιγότερο ειδική. Εθνική ταυτότητα ακόμα πιο γενική. Και η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι μια φαρδιά ομπρέλα που χωράει όλου. Δεν μπορώ να σα δώσω έναν πολύ συγκεκριμένο ορισμό της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Νομίζω όμως ότι τα πολύ θεμελιώδη φαινόμενα της ζωής δεν είναι εύκολο να οριστούν. Δεν μπορεί να οριστεί η ζωή, δεν μπορεί να οριστεί ο θάνατος, δεν μπορούμε να ορίσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την αισθάνεται κανείς όμως. Διότι συναισθανόμαστε ένα είδος αλληλεγγύης ημέν προς τους δε. Όταν βλέπουμε ένα κτίριο στην Ελλάδα για παράδειγμα, αισθανόμαστε μια οικειότητα. Έχουμε και τους ήρωες της ευρωπαϊκής ταυτότητας που δεν είναι πλέον, ο Αριστοτέλης για παράδειγμα, δεν μονάχα Έλληνας, είναι όλων των Ευρωπαίων. Έχουμε προσωπικότητες, έχουμε ήρωες, έχουμε μνημεία, Έχουμε μνημεία απτά αλλά και άειλα και η αρχαία πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι πια μονάχα των Ελλήνων, είναι η κοινή πολιτιστική κληρονομιά των Ευρωπαίων. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία συναποτελούν την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα θα είναι πραγματικά συμπεριληπτική. Θα του περιλαμβάνει όλου. δηλαδή, αλλά χρειαζόμαστε μια στέρεα αραχοκοκαλιά και αυτή είναι η κοινή μας κληρονομιά. Και γι' αυτό το έτος ευρωπαϊκής κληρονομιάς είναι πολύ σημαντικό. Οι δυσκολίες για την ανάπτυξη της παιδείας βεβαίως. Λιτότητα, περικοπές στις ε, δαπάνες της παιδείας. Δυστυχώς η Ευρώπη υστερεί, η Ασία την ξεπερνά, η Αμερική επίσης. Η Αμερική και η Ασία επενδύουν πολύ περισσότερα από εμάς τονίζουμε διαρκώς την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων αλλά και ευφιέστερων επενδύσεων στην παιδεία. Διότι περισσότερα χρήματα από μόνα του δεν αρκούν. Πρέπει να επενδύσουμε με ευφιέστερο τρόπο στην παιδεία. Και γι' αυτό στη διάσκεψη κορυφή για την παιδεία ένα από τα βασικότερα θα είναι οι ευφυεί επενδύσει, Όχι μόνο για τα ενδιαφερόμενα μέρη τα δικά μα, αλλά και με υπουργούς και από άλλους τομείς αρμοδιότητας για τις βασικές δεξιότητες, όχι μόνο, ασφαλώς όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες, που οι τεχνικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές, αλλά, αναφερθώ και στη δική σας παρέμβαση, δείχνει προς την κυρία Μπίλτ, έχουμε σημαντικές δυσκολίες με τις βασικές κοινωνικές ε, δεξιότητες, για παράδειγμα αλφαβητισμό και χρήση της αριθμητικής σε πολλές χώρες έχουμε σημαντικά προβλήματα αλφαβητισμού και πολλοί έχουν προβλήματα με τη σωστή χρήση της αριθμητικής. Βασικά πράγματα δηλαδή. Τα σχολεία οφείλουν να διδάσκουν αυτά τα βασικά, τα θεμελιώδη πράγματα. Οι τεχνικές, οι ψηφιακές δεξιότητες θα πρέπει να έρθουν μετά, αφού θα έχουν διδαχτεί τα παιδιά όλα αυτά τα παραδοσιακά, αλλά και τις κοινωνικές δεξιότητες, διότι θεωρώ ότι λόγω των αλλαγών που επισυμβαίνουν στην κοινωνία το σχολείο καλείται να διδάξει στο παιδί πώς θα ζήσει μέσα σε μια κοινότητα, πώς θα συζητήσει, με, θα συνομιλήσει με τα άλλα μέλη της ομάδας, πώς θα αντιμετωπίσει περίπλοκες καταστάσεις και ούτω καθεξής. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να διδάξει κάποιες βασικές θεμελιώδεις κοινωνικές δεξιότητες που συνήθως τα αναλαμβάνουν αυτά οι οικογένειες, αλλά δυστυχώς τώρα τα σχολεία καλούνται νομίζω να παίξουν σημαντικότερο ρόλο στην διδασκαλία αυτών των δεξιοτήτων. Τώρα για την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Κοιτάξτε, τώρα εμείς εργαζόμαστε για να συνδυάσουμε τον έρασμο χωρίς χαρτιά, άμρακ και την ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα με ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων των φοιτητών μεταξύ των συμμετεχών των πανεπιστημίων με στόχο να ενισχυθούν τα προγράμματα αυτά και να επιτρέπεται σε Ευρωπαίους φοιτητές να μπορούν να σπουδάζουν σε άλλες χώρες και να μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους με ευκολότερο τρόπο. Η λύση αυτή θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις ε, χώρες μέλη με ένα ενιαίο κώδικα, κωδικό αριθμό δηλαδή, με μια ενιαία ταυτότητα και με ηλεκτρονικό τρόπο μετάδοσης των δεδομένων. Αυτό σε όλα τα προγράμματα έρασμος και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική κάρτα ταυτότητας στην βάση του συστήματος EIDS. Και τέλος η στρατηγική για τον πολιτισμό και τον ψηφιακό κόσμο συνδυάζει τα δύο αυτά. Έχει έξι αντικειμενικούς στόχους. Πρώτος, διασφάλιση ευρύτερης και δημοκρατικότερης πρόσβαση στον πολιτισμό. Δεύτερο, προώθηση, μάρκετινγκ και αξιολόγηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενδυνάμωση της ψηφιακής παραγωγικότητας. Πέμπτο, οι μικρές και μισές επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτά να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τέλος ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας. Και τέλος η ενίσχυση του παραδοσιακού τμήματος της Creative Europe. Γνωρίζετε ότι λόγω της ιδιαίτερης πολιτικής μας κατάστασης το 2014 είχαμε τις δυσκολίε που είχαμε. Ελπίζω στο μέλλον και μάλιστα ο επόμενος επίτροπος θα συμβάλλει στην προσπάθεια τη δική σας να παντρέψετε τα δυο αυτά μέρη της ε, ε, Creative Europe. Ε, ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Ε, θεωρώ ότι τα δύο μέρη, θεώρησα διαβάζοντας το κείμενο της Κομισιόν ότι τα δύο μέρη του προγράμματος θα ξεχωρίζονταν, θα διαχωρίζονταν πάλι. Αλλά αν είναι διαφορετικά δεν έχουμε πρόβλημα. Ε, πολλές ε, ήταν οι ερωτήσεις και έπρεπε να απαντηθούν ε, διεξοδικά με τον Επίτροπο. Προχωρούμε στον επόμενο γύρο και θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Λοιπόν, αυτά είναι τα ονόματα των συμμετεχόντων στο δεύτερο γύρο. Ένα λεπτό, παρακαλώ, να μιλήσετε για να προλάβει να απαντήσει και ο Επίτροπος. Ο κύριος Στογεύσκη. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για το Brexit. Οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν πολύ αλλά είναι πολύ σημαντικές σε σχέση με το Erasmus Plus. Η παιδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ελκυστική για τους Ευρωπαίους και έχουμε πολλούς σπουδαστές που χρησιμοποιούν το Erasmus Plus στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πιο πολύ από ότι αντίστροφα. Ερώτηση. Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου εδώ. Πώς μπορεί ενδεχομένως να εξασφαλιστεί μια συνέχεια αυτών των προγραμμάτων και ε, συνέχεια των συνεισφορών επίσης. Δεύτερη ερώτηση. Έχουμε πολλές ε, συμφωνίες ε, με το Ηνωμένο Βασίλειο, ασφάλιση εργοτέχνης κλπ. Υπάρχει περίπτωση στο τέλος των διαπραγματεύσεων για τον Brexit να υπάρξει κάποια βεβαιότητα ώστε να συνεχιστούν οι συμβάσεις, οι συμφωνίες που υπάρχουν στον τομέα του πολιτισμού. Η Ευχαριστώ πολύ. Να πω μόνο ότι απογοητεύτηκα που οι έξι προτάσει, κύριες προτάσεις πολιτικής από την δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένε διατάξεις για να κάνουμε δράσεις σε επίπεδο βάση σε επίπεδο πολιτών. Για τους καλλιτέχνε α πούμε, που είναι νέοι, ώστε να πειραματιστούν και να ρηψοκινδυνεύσουν. Θα ήθελα να προτείνω με έχοντας κατά νου τα χρόνια της χρονής κουλτούρας που έχουμε μπροστά μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το ένδοξο παρελθόν μας, πολιτιστικό παρελθόν μας και μάλιστα ιδιαίτερα τη στιγμή που διάφορες κοινότητες διαφοροποιημένες δέχονται μεγάλες πιέσεις λόγω ισλαμοφοβίας και άλλων παραγόντων. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα πρέπει να βασιζόμαστε μόνο στην χριστιανο-ιουδαϊκή παράδοση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Γιατί οι μεγάλες ανακαλύψεις στα μαθηματικά, στην επιστήμη, στην αστρονομία προέρχονταν από άλλους πολιτισμούς, από τους Άραβες ας πούμε. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν και τον Επίτροπο να δει και το χίλιες και μία εφευρέσεις που κάνουν πολλή δουλειά σε αυτό το πράγμα και για τους νέους και το Brexit. Κάποιοι είναι εξοργισμένοι και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εδώ σήμερα και θέλουν ακριβώς οι, οι εκπρόσωποι τους εδώ στο Κοινοβούλιο να κάνουν κάτι για αυτούς. Κυρία Σιόρντοβα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Επίτροπο για την παρουσίαση. Εγώ έχω μια πληροφορία να σας δώσω για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Συζητάμε τον κανονισμό του, όπως ξέρετε, και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε γρήγορα με τις εκθέσεις. Έχουμε γύρω στις 200 τροπολογίες και νομίζω ότι υπάρχουν δύο κύρια σημεία εδώ. Καταρχάς το να έχουμε νέα κονδύλια για αυτά τα προγράμματα, αυτά τα νέα προγράμματα και κατά δεύτερον λόγο, δεν θέλουμε να χάσουμε ή να παραβλέψουμε αυτά που έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Εθελοντισμού. Να μην ξεχνάμε λοιπόν τι έχει πετύχει ο εθελοντισμός, τι στόχους έχει και τι αξίες έχει στα πλαίσια του νέου προγράμματος. Όπως επίσης και στην ονοματοδοσία που θα κάνουμε αυτό του νέου προγράμματος. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καλή συνεργασία και να υπάρχει μια καλή σχέση στις διαπραγματεύσεις που θα έχουμε με την Κομισιόν και τη Συμβουλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Βέντα. Ευχαριστώ πολύ. Χθες δόθηκαν, απονεμήθηκαν τα πρώτα ε, βραβεία ε, στα πλαίσια του προγράμματός σας η Κομισιόν πώς θα στηρίξει άτομα με αναπηρία στον τομέα του αθλητισμού. Ε, εγώ ασχολήθηκα και με το θέμα του στισίματος των αγώνων που είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να ε, ισχύσει η συμφωνία για το στήσιμο των αγώνων. Είχαν γίνει πολλές ε, ανακοινώσεις σε αυτόν τον τομέα από τότε και μετά. Τι έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νίκοφ. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με την αναγνώριση συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα στα πλαίσια των συμφωνιών για την αναγνώριση συμμετοχής αλληλεγγύης έχετε πρόθεση να αναγνωρίσετε τη συμμετοχή αυτή ως μορφή δεξιότητας άτυπης στα πλαίσια λοιπόν του της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού προβλέπεται και ύπαρξη ενός πάσου, ενός ελευθέρας. Μήπως αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για την κινητικότητα των νέων. Νομίζω ότι τα κριτήρια αξιολόγησης αυτής της νέας πρωτοβουλίας περιλαμβάνουν ε, κριτήρια ποσοτικά εις βάρος των ποιοτικών κριτήριων. Αυτά ευχαριστώ. Κύριε Σαμίτ, Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα. Είναι βέβαιο ότι η πολιτιστική μας κληρονομιά αποτελεί ένα το κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Στη Μάλτα αυτό το ζούμε ιδιαίτερα γιατί η πρωτεύουσά μας η Βαλέτα θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και αυτό συμπίπτει και με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού. Τώρα το ερώτημά μου είναι το εξής. Εκτίμησα πολύ τις αναφορές που κάνατε στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Μιλήσατε και για τα ΜΜΕ και την γνώση ώστε να καταπολεμήσουμε τις ψευτικές ειδήσει. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα, νέες μεθόδους για νέα ψηφιακά συστήματα ενδεχομένως. Και κάτι άλλο, μια ερώτηση. Πώς προετοιμάζεται η Κομισιόν για τα τεράστια άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα πρέπει να διδάξουμε τις αξίες μας για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να περιλαμβάνονται αυτά στην ταυτότητά μας. Θα πρέπει να, τα περιλάβουμε όλα αυτά στα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Γιατί αυτές ακριβώς τις αξίες δεν τις τονίζουμε, δεν, την, δεν τις υπογραμμίζουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δυστυχώ θα καταστήσουμε καινή γράμματο όλη την εκπαίδευσή μα. Και άψυχη, ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία, κυρία Λιμπέρτσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση και για τις ε, ανακοινώσεις σας που είναι σημαντικές. Φαίνεται ότι το θέμα της παιδείας είναι πολύ σημαντικό, γίνεται σημαντικό. Τρεις ερωτήσεις. Χαίρομαι που είπατε ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο συμμετεχόντων και να συμπεριλάβουμε και τους, ε, τα μειονεκτικά άτομα. Ε, είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρξει όντως χρηματοδότηση η προσαρμογή των ε, κονδυλίων θα πρέπει να αυξηθούν για να λάβουν υπόψη την αύξηση του κόστου ζωής στο, στη χώρα υποδοχής. Ένα άλλο σημαντικό είναι να δώσουμε έμφαση στο διδακτικό προσωπικό ε, που είναι απαραίτητο για όλα αυτά. Επίσης, ε, άτυπη διαβίου μάθηση ε, είναι ένας τομέας που πρέπει να προωθηθεί ακόμα περισσότερο. Τέλος, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Χώρου. Μετά την Πολόνια θα πρέπει να δοθεί συνέχεια. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάποια συγκεκριμένα βήματα έχουν γίνει για την αμοιβαία αναγνώριση των πανεπιστημίων, της ισοτιμίας και των δεξιοτήτων. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και το χαιρετίζω επίσης να πω και το εξής. Η Κομισιόν φαίνεται ότι έχει θέσει ένα εκπαιδευτικό στόχο μέχρι το 2025 να μιλούν φοιτητέ δύο επιπλέον ξένες γλώσσε, πέραν τη μητρική δηλαδή. Αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα για τι μειονότητε. Και νομίζω ότι αποτελεί στην ουσία την βάση για συνύπαρξη και συνεργασία. Το γεγονός ότι δηλαδή ο ένας μιλά τη γλώσσα του άλλου. Έχω μια ερώτηση, την εξή. Και οι χώρε της Ανατολική εταιρική σχέση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα πλαίσια αυτών των προγραμμάτων. Οπότε η συμμετοχή του ακριβώ με ποιο τρόπο θα ελοπίθει. Ευχαριστώ. Περίμενα τη μετάφραση μέχρι να τελειώσει. Ο συνάλφος Βέρτ, τελευταίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισήγησή σας. Νομίζω ότι έχετε το καλύτερο χαρτοφυλάκιο στην Κομισιόν. Να μην πολύ μιλήσω για το Erasmus Συν, αλλά διάβασα την έκθεση και τη μελέτη και βλέπω ότι η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με λογισμικό το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα θεσμικά μάλλον στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η ανοιχτή ηλεκτρονική πόρη στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι μελλοντικά αυτή οι ψηφιακή πόροι θα έχουν τεράστια σημασία Δηλαδή θα είναι πολύ πιο σημαντική από του παραδοσιακού πόρους σε αυτό τον τομέα. Νομίζω λοιπόν είναι σημαντικό που η Κομισιόν έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να δημιουργήσουμε ψηφιακές πλατφόρμες οι οποίες θα είναι διαθέσιμε στους τελικούς χρήστες δωρεάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ξανά έχετε το λόγο για να απαντήσετε στις πολλές ερωτήσεις που μας απασχολούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να πω για το Brexit. Έχουμε ενεξελίξει διαπραγματεύσεις, ακόμα δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα καταλήξουν, τι θα προκύψει. Μέχρι το τέλος των διαπραγματεύσεων λοιπόν, όπως αναφέρει η συνθήκη, έχει πλήρη δικαιώματα, πλήρες μέλος δηλαδή, το Ενωμένο Βασίλειο. Ε, Συμμετέχει δηλαδή στο Εράσμους ΣΥΝ και μπορεί να χρησιμοποιήσει Κανεί τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να σπουδάσει στο Ενωμένο Βασίλειο χάρη σε αυτό. Μέχρι να αποχωρήσει πλήρως το Ενωμένο Βασίλειο από την Ένωση. Θα δούμε πώ θα καταλήξουν οι πραγματεύσεις. λοιπόν. Τώρα για το κόπηρα, τα πνευματικά δικαιώματα. Σωστή ερώτηση. Τι θα γίνει αφού εφαρμοστεί από ό,τι ξέρω υπάρχουν γύρω στις χίλιες τροπολογίες για αυτό το θέμα από το Κοινοβούλιο. Οπότε δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα πάμε. Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Είναι πολύ αργή η διαδικασία. Είναι περίπλοκη. Οπότε να δούμε. Θα περιμένουμε αναγκαστικά αλλά η ασφάλεια δικαίου θα υπάρχει όπως υπάρχει και σε άλλες περιπτώσεις. Θα υπάρχει δηλαδή όλος αυτός ο μηχανισμός ο οποίος διασφαλίζει την νομική ασφάλεια για τη νέα κατάσταση. Αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, προς το παρόν τουλάχιστον. για τις δράσεις σε επίπεδο βάσης πολιτών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι να σας πω ότι η Ευρώπη αποτελεί το μεγαλύτερο παράγοντα χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων σε επίπεδο βάσης. Ας πούμε στον αθλητισμό. Έχουμε όμως και την υποχρέωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών να κάνουν κάτι. Εμείς βεβαίως παρέχουμε κάποια χρηματοδότηση, κάποια υποστήριξη, αλλά αυτό αποτελεί, μάλλον διοχετεύεται μέσω μιας συμπληρωματικής σημαντικής βοήθειας ή μέσω, την παροχή ενός, μέσω της παροχής ενός πλαισίου Βεβαίω μπορούν να χρηματοδοτηθούν και διασυνοριακές μορφές που παρουσιάζουν δηλαδή ευρωπαϊκή διάσταση. Ξέρετε αυτό είναι πάντοτε το πρόβλημα με τα μικρής κλίμακας προγράμματα ότι η Ευρώπη είναι υπερβολικά μεγάλη για αυτά τα μικρά προγράμματα. Δηλαδή χρηματοδοτούν συζητούμε κάποιες μορφές συνεργασίας όπως τις διασυνοριακές αλλά νομίζω ότι ο ρόλος της χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων και των παρεμβάσεων σε επίπεδο βάσης νομίζω εμπίπτει περισσότερο σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές. Οπωσδήποτε δεν θα ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αποκλεί κάποια πράγματα. Ας πούμε, αποκλεί επιρροές και διαδράσεις με άλλους πολιτισμούς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τη Βοσνία στην Ευρώπη, όπου έχουμε μια κοινότητα μουσουλμάνων, που δεν είναι μόνο μια σημαντική κοινότητα σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι μια κοινότητα που είναι σημαντική σε διεθνές πολιτιστικό επίπεδο. Υπάρχει εδώ και μισή χιλιετία. Είναι λοιπόν σημαντικό για τους Βόσνιου αλλά και για τους Κοράτες να περιλάβουν την Ισλαμική επιρροή στην Ιουδοχριστιανική ε, πολιτιστική τους ε, σκοπιά. Μπορούμε να, έχουμε, να έχουμε λοιπόν μια διάδραση με την, σε σχέση με την επιρροή που είχαν άλλοι πολιτισμοί στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Και θα ήθελα πραγματικά να υπάρχει μια ευκαιρία για τις τοπικές κοινότητες να, αντιμετω... να έρθουν ενώπιον στον οποίο, με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, με την πολιτιστική τους κληρονομιά. Για να κατανοήσουν δηλαδή πόσο σημαντική είναι αυτή η διάδραση με τους όλους πολιτισμούς και να συζητήσουμε βεβαίω όλα τα απτά και μη στοιχεία αυτής της δικής τους πολιτιστικής κληρονομιάς. Και για τους νέους τώρα που είναι εξοργισμένοι με τον Brexit, τι να σας πω, απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αυτή, δεν ήταν δικιά μας, τους καταλαβαίνω, είναι εξοργισμένοι. Και κάποιοι από εμά το ίδιο, αλλά ήταν νόμιμη, θεμητή απόφαση αυτή. Ναι, και όχι μόνο οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι. Ναι, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχουν και κάποιοι, όχι και τόσο νέοι, που είναι εξίσου εξοργισμένοι με την Βρετανική απόφαση για τον Brexit. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η κατάσταση. Uh, how to support disabled people. Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό. Έχουμε κάποια προγράμματα στα πλαίσια του Erasmus Plus για αθλητικές δραστηριότητες σε επίπεδο συλλόγων με στόχο την κοινωνική ένταξη αυτών των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε ας πούμε αυτό το βραβείο βραβεία που παρέδωσα χθε το βράδυ, τρία κιόλα. Το ένα από αυτά τα βραβεία αφορούσε συγκεκριμένα την ένταξη ατόμων με αναπηρία ώστε ακριβώς να έχουν μια ουσιώδη και ενεργό ζωή στα πλαίσια του αθλητισμού. Δυστυχώς δεν έχω κάτι άλλο νέο ω στοιχείο να σας δώσω εδώ. Το θέμα βρίσκεται ακόμα στο Συμβούλιο και για την χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή 45 οργανώσεις που έχουν υπογράψει αυτή την κοινή δήλωση και συνεχώς καλούμε νέες οργανώσεις και άλλες οργανώσεις να προσυπογράψουν αυτή τη δήλωση, αυτή την κοινή δήλωση. Τα κριτήρια για το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Σώμα είναι ακριβώς τα ίδια με τα κριτήρια για, το, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού. Το σώμα βέβαια θα έχει δικό του χωριστό κονδύλι, προπολογισμό. Και νομίζω ότι για το μέλλον μπορεί να δώσει περισσότερη έτσι, σταθερότητα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού στο παρελθόν ώστε να υπάρχει μια πιο στέρεη βάση για όλους με περισσότερα χρήματα και κυρίως για τους ίδιους τους εθελοντές. Τώρα, η αξιοποίηση της ε, τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας για την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην ε, εκπαίδευση. Ε, ετοιμάζουμε μια ανακοίνωση κιόλα από αυτού για την αξία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, γιατί οι καιροί πραγματικά είναι πονηρή. Αν θέλουμε να έχουμε μια πιο συνεκτική κοινωνία στην Ευρώπη και να έχουμε μια κοινωνία έτοιμη θα πρέπει να βασιζόμαστε στις κοινέ μας ε, αξίες. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα δύσκολο ζήτημα, περίπλοκο. Εξελίσσεται συνεχώς, υπάρχουν καινοτομίες ε, και υπάρχει και η αντίστοιχη εκπαίδευση που προσπαθεί να ακολουθήσει τον βηματισμό της εξέλιξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Αλλά νομίζω ότι εδώ ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι η έλλειψη ευελιξίας των εκπαιδευτικών συστημάτων και αυτό ακριβώς στοχεύουμε στο να κάνουμε τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο ελαστικά ώστε να επιτρέπουν στους νέους να αυτοπροσαρμόζονται στην εξέλιξη των καινοτομιών. Για τα εκπαιδευτικά μειονεκτήματα και το Erasmus Sin. Γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε αύξηση των κοντιλίων στο Erasmus Sin για να διευρύνουμε το πεδίο και να, να περιλάβουμε ε, μειονεκτούσες ομάδες στο Erasmus Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπατε. Είναι πολύ σημαντικό το Erasmus για την κινητικότητα των νέων και των φοιτητών. γιατί πραγματικά βοηθούν στο να προσεγγίσουμε την Ευρώπη ως μια κοινή οικογένεια. Θα έχουμε μια υπουργική συνάντηση το Μάη στο Παρίσι και αυτό θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία καταγραφής της πραγματικότητας. Ο ευρωπαϊκός εκπαιδευτικός χώρος τώρα δυστυχώς περιορίζεται προς το παρόν στις χώρες ΕΕ αλλά το γεωργικό πεδίο του Εράσμου πηγαίνει πέραν των χωρών της Ένωσης. Οπότε και εδώ έχουμε ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο προς αυτήν Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά κύριε Επίτροπε που σήμερα μας ενημερώσατε, μας απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε θα μας απασχολούν συνέχεια μέχρι το τέλος της θητείας μας. Θα κάνουμε πολλές συζητήσεις και για το Erasmus Plus και για το πρόγραμμα Creative Europe και για την πρικοδότησή τους. Και σε αυτό το σημείο Θέλω να επαναλάβω την ε, διακαή μας επιθυμία και κατεπίγουσα παράκληση οι προτάσεις για το μέλλον των προγραμμάτων να ε, δοθούν σε μας το ταχύτερο δυνατόν για να προλάβουμε και εμείς μέσα σε αυτή τη θητεία ως Κοινοβούλιο να κάνουμε την πρώτη δουλειά, να κάνουμε την πρώτη ανάγνωση, ούτως ώστε το επόμενο Κοινοβούλιο να μην χρειαστεί να θα αρχίσει όλα από την αρχή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Ο κύριο Επίτροπος Έτιγκερ συνεννοήθηκε με το Κοινοβούλιο ότι τα στοιχεία θα δοθούν το Μάιο. Παρ' όλα αυτά, την περασμένη φορά κάναμε διαπραγματεύσεις μέχρι τέλους πάλι χωρίς νούμερα και στοιχεία. Ε, σημασία έχει και η δομή των προγραμμάτων στο Creative Europe. Μπορούμε να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε στο Erasmus Plus, ποια τμήματα θα έχει, τι ποσοστό θα έχει το κάθε τμήμα, τι στόχο θα εξυπηρετεί το κάθε τμήμα. Υπάρχουν θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα νούμερα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, θερμή παράκληση, δώστε μας το ταχύτερο δυνατόν τα προγράμματα, ε, ακόμα κι αν δεν υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία στα πλαίσια του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα μας βοηθήσει αυτό να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, με, υπευθυνότητα. Να μην αφήσουμε μια κληρονομιά κακή στο επόμενο κοινοβούλιο όπου θα αναγκαστούν να ξαναρχίσουν από την αρχή. Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιερώσατε. Θα παραμείνουμε σε επικοδομητικό και κριτικό διάλογο, όπως λέγεται έτσι τόσο ωραία, και χαίρομαι για την περαιτέρω συνεργασία με εσάς και την ομάδα σας. Ευχαριστώ.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 Uh, Θα περιμένουμε λίγα λεπτά να επιστρέψουν κάποια μέλη. Και φαίνεται χρειάστηκαν ένα μικρό διάλειμμα. Γιατί είχαμε και προηγούμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλώς ορίζω όλους στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνεδρίασης. Ελπίζω ότι τα μέλη που έφυγαν θα επανέλθουν. Έτσι είπαν τουλάχιστον. Όπως ξέρετε, ο πρόεδρος Σταγιάννη με την υποστήριξη της διάσκεψης των πρόεδρων πρότεινε αυτή τη βδομάδα να οργανωθεί εδώ στο Κοινοβούλιο μια Αφρικανική εβδομάδα ούτως ώστε να αναδειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής Αφρική Ευρωπαϊκή Ένωση του Αμπιτζάν 29 και 30 Νοεμβρίου. Όλες οι επιτροπές εκλήθησαν να συμμετάσχουν σε αυτή την Αφρικανική εβδομάδα και έτσι αυτή τη βδομάδα ε, εστίασαν στις συνεδριάσεις τους σε ένα ειδικό θέμα σε ένα ειδικό σημείο από το θέμα σχέσης ε, Ένωσης Αφρικής. Εμείς ε, ασχοληθήκαμε ε, αναδεικνύοντας την πολιτική συμμετοχή των νέων, ε, την παιδεία, τον πολιτισμό. Ε, θα ακούσουμε σήμερα ομιλίες από την Επιτροπή την UNESCO, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νέων και από, θα ακούσουμε και Αφρικανούς εκπροσώπους. Πριν δώσω το λόγο στη, στον πρώτο ομιλητή, θα ήθελα να καλωσορίσω ε, ιδιαίτερους προσκεκλημένους, μια αντιπροσωπεία του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, που είναι οι φιλοξενούμενοι μας αυτή τη βδομάδα και μια αντιπροσωπεία από την Εθνοσυνέλευση της Νιγερίας. Χαίρομαι πολύ που ήρθατε σήμερα και είστε εδώ και ελπίζω ότι η συζήτησή μας θα είναι και για τη δική σας τη δουλειά χρήσιμη. Θα αρχίσω με ανταλλαγή απόψεων με παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μορέλ είναι ε, επικεφαλής του τμήματος ε, της Γενικής Διεύθυνσης ε, εκπαίδευση και Πολιτισμού για τη Διεθνή Συνεργασία και θα μας παρουσιάσει τα, τις νέες προσπάθειες που γίνονται στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης Αφρική-Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ό,τι 10 λεπτά και μετά θα παρουσιάσουμε και τους άλλους ομιλητές. Η κυρία Μορέλ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την ευκαιρία που μου δίνετε να εξηγήσω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της συνεργασίας για την παιδεία με την Αφρική. Η συνεργασία αυτή δεν είναι βεβαίως νέα. Συνεργαζόμαστε με την Αφρική ε, εδώ και πολλές δεκαετίες. Θα μιλήσω ιδιαίτερα για τον ρόλο που παίζει η Αφρική στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus δηλαδή θα μιλήσουμε κυρίως για ανώτερη εκπαίδευση, αλλά θα εξηγήσω ακόμη τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να αρχίσουμε λοιπόν υπενθυμίζοντάς σας ότι οι προτεραιότητές μας είναι, όπως θα δείτε, τους διάφορους τομείς στην διαφάνεια, διασυνδέονται Θέλουμε δηλαδή να ενισχύσουμε πρώτα την διακυβέρνηση στην Αφρική με ισχυρό κράτος δικαίου. Θέλουμε να εργαστούμε για την πρόληψη συγκρούσεων και να αντιμετωπίζουμε κρίσεις πριν να λάβουν χώρα. Να εργαστούμε για την βιώσιμη ανάπτυξη. Να συνεργαστούμε για την κινητικότητα και μετανάστευση. Χρειαζόμαστε ανθρώπους εκεί με γερή παιδεία και όλοι αυτοί οι στόχοι είναι απολύτως αλληλοσυνδεδεμένοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μεγαλύτερος δωρητής στον χώρο της παιδείας στην Αφρική με καλύτερη στήριξη για πολλές αφρικανικές χώρες. Για την ώρα 29 αφρικανικές χώρες έχουν θέσει την παιδεία ως πρώτη στην προτεραιότητά τους σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει ή σχεδιάζει να επενδύσει σχεδόν 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την παρούσα ε, προγραμματική περίοδο για να στηρίξει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδίως μεταξύ ε, ε, μη προνομιούχων νέων, νέων με αναπηρίες, ιδίως για τα κόριτσια, για ε, μειονότητες, διότι οι περισσότεροι νεαροί Αφρικανοί δεν ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όταν το καταφέρνουν δεν αποκτούν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες. Εκτός από την καλύτερη στήριξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει σημαντικά διάφορες πρωτοβουλίες όπως ε, την Global Partnership for Education της Παγκόσμιας Τράπεζας, άλλη ε, πρωτοβουλία για ε, εκτοπισμένους και για πρόσφυγες εντός Αφρικής. Θα ήθελα τώρα να έλθουμε ιδίως στο πρόγραμμα Erasmus διότι η Αφρική από την αρχή της παρούσας προγραμματικής περίοδου είναι σημαντικός εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus Να σας εξηγήσω τι κάνουμε στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης μέσα στα πλαίσια του Erasmus Έχουμε διάφορους τρόπους για να, για να επιτρέψουμε την εμπλοκή των Αφρικανικών Πανεπιστημίων. Νομίζουμε ότι είναι σημαντικό τα Αφρικανικά Πανεπιστήμια να ενταχθούν στα διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και δίκτυα ερευνητών να μην μείνουν εκτός των δικτύων αυτών και θεωρούμε ότι ο Erasmus είναι ένα σημαντικός μηχανισμός που επιτρέπει στα Αφρικανικά πανεπιστήμια να εντάσσονται στα δίκτυα αυτά. Και υπάρχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο από την Αφρική αλλά και από την Ευρώπη για συνεργασία με Αφρικανικές χώρε. Για την ώρα η ιδέα είναι ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση, να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα των Αφρικανικών πανεπιστήμιων εξελίσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προσφέρουν υψηλότερη ποιότητα και είναι πιο προσαρμοσμένα στις ανάγκες ε, της αγοράς και ε, της ε, κοινωνίας γενικότερα. Η παραδοσιακή κινητικότητα έρασμος που γνωρίζουμε στην Ευρώπη άνοιξε για όλο τον κόσμο το 2014 και επομένως και για την Αφρική και από το 2015 μπορέσαμε να χρηματοδοτήσουμε 10.000 ε, κινήσεις ε, και φοιτητών και καθηγητών και άλλου διδακτικού προσωπικού από την ε, Αφρική να έρθουν στην Ευρώπη και επίσης να πάνε μεταπτυχιακοί φοιτητές δικοί μας στην Αφρική. Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε μέχρι δηλαδή της προγραμματικής περίοδου να διπλασιάσουμε τον αριθμό αυτό. Εκτός του Erasmus που αναφέρεται ιδίως στην κινητικότητα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, έχουμε και ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της κινητικότητας ενδοαφρικανικά, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της κινητικότητας εντός της Αφρικής, διότι οι αφρικανικές χώρες μας λένε ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουν δείκτε συνεργασία με την Ευρώπη, αλλά ε, επιθυμούν να αναπτύξουν και τη συνεργασία μεταξύ τους. Με βάση αυτή την, αυτά τα προγράμματα κινητικότητα εντό Αφρικής μπορέσαμε να ε, υποστηρίξουμε πάνω από 800, 800 φοιτητές και περίπου 200 εκπαιδευτικούς με υποτροφίες Εράσμους Μούντους για φοιτητές και Εκτός της κινητικότητας, στα πλαίσια του Ερασμοσύν, προσφέρουμε και χρηματοδότηση για capacity building, για να επιτρέψουμε δηλαδή σε αφρικανικά πανεπιστήμια να συνεργαστούν με ευρωπαϊκά. Εκτός από την συνεργασία αυτή στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης, υπάρχει και μια πτυχή νεότητας στο πρόγραμμα Erasmus, όπου οι νέοι και οι νέες έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται σε project capacity building και όχι μόνο οι νέοι και οι νέες αλλά και οργανώσεις νέων. Εργαζόμαστε και ε, ε, ε, επί ενός tuning project όπως το αποκαλούμε για την εναρμόνιση των συστημάτων ανώτερης εκπαίδευσης στην Αφρική και όχι μόνο στην Αφρική αλλά και σε συνεργασία με την Ευρώπη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε κοινά συστήματα βαθμών credit που θα λειτουργήσουν μέσα στην Αφρική και θα επιτρέψουν καλύτερη ε, αναγνώριση των προσόντων και επομένως κινητικότητα και με την Ευρώπη γιατί ε, πάσχουν τα συστήματα από έλλειψη συγκρισιμότητας. Μέσα στο Tuning Project λοιπόν εργαζόμεθα επίσης και για την εναρμόνιση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, ώστε οι αφρικανικές χώρες να έχουν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη η μια στα εκπαιδευτικά συστήματα της άλλης και αυτό να ενισχύσει πάλι με τη σειρά του την κινητικότητα. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια για την ε, ενίσχυση των ερευνητών. Για την ώρα η Αφρική δεν συμμετέχει πάρα πολύ. Από την αρχή της παρούσας προγραμματικής περίοδου έχουμε χρηματοδοτήσει μονάχα 500 Αφρικανούς ερευνητές. Υπάρχει όμως πολύ ενδιαφέρον και προθυμία από την πλευρά Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ιδρυμάτων να προωθηθεί αυτή η συνεργασία, δηλαδή να ενταθεί η κινητικότητα των ερευνητών σε όλες τις φάσεις της σταδιοδρομίας τους. Για την ανανεωμένη συνεργασία με την Αφρική υπάρχουν τρεις εμβληματικέ πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε προτείνει στην Αφρικανική Ένωση και θα τα συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα στην διάσκεψη κορυφή. Το πρώτο είναι ένα πρόγραμμα για την ενδυνάμωση της νεολαία, ένα είδος επέκτασης της πρωτοβουλίας νεολαία του Έρασμο ΣΥΝ που στοχεύει στην ε, στήριξη οργανώσεων βάσης να ενταχθούν σε project κινητικότητα και να βελτιώσουν την διακυβέρνησή τους. Δεύτερη εμβληματική πρωτοβουλία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την κινητικότητα στα πλαίσια τη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Για την ώρα η κινητικότητα περιορίζεται στην ανώτατη εκπαίδευση, γι' αυτό θέλουμε να περιλάβουμε σε αυτήν και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να ενισχύσουμε το αφρικανικό κεφάλαιο των ε, ε, ενώσεων αποφύτων μας, ώστε οι φοιτητέ μας όταν είναι στην Ευρώπη να μπορούν να συνεχίσουν ενώ άλλοι φοιτητέ και νέοι ερευνητέ να επιστρέψουν στην Αφρική. Αυτό όμως να επιτρέψει μια μακρά πνοή συνεργασία με την Αφρική. Έχουμε διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις μέχρι τη διάσκεψη κορυφής και τον διαρθωμένο διάλογο με φοιτητέ και αποφύτους Φοιτητέ και απόφοιτοι έχουν απευθύνει έκκληση στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων που θα συνέλθουν την επόμενη εβδομάδα, ιδίω ζητώντα εναρμόνιση. Θέλουν εναρμόνιση των συστημάτων ανώτερη εκπαίδευση που θα του επιτρέψουν να ε, ε, διατηρήσουν μια κινητικότητα όχι μόνο με την Ευρώπη αλλά και εντό τη Αφρική. Και όταν θα αναλάβουν εργασία, όταν θα μπουν στην παραγωγή πλέον, να μπορούν να είναι κινητικοί και εντό Αφρική. από την ε, Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ είχα προβλέψει συναδέλφους οι οποίοι θα σας έλεγαν και άλλα πράγματα αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συνεργασία για τα πολιτιστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει έναν αριθμό project στον τομέα του πολιτισμού διότι θεωρούμε ότι οι δημιουργικές βιομηχανίες εντό εισαγωγικών μπορούν να έχουν σημαντική θετική επίπτωση στην απασχόληση, να δημιουργήσουν πολλές δουλειέ για τους νέους στην Αφρική Βλέπουμε επίσης ότι στον τομέα του πολιτισμού παίζουν σημαντικό ρόλο οι γυναίκες. Είναι ένας τομέας όπου ο ρόλος των γυναικών είναι ζωτικός. Και των γυναικών και των νέων. Εδώ λοιπόν αναπτύσσεται ένα αριθμός πρωτοβουλειών τις οποίες χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα συνεχίσει να τις χρηματοδοτεί και θα ήθελα επίσης να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό πρόγραμμα Inter-ACP, εντός δηλαδή των χώρων ΑΚΕ. Θα αρκεστώ σε αυτά τα λόγια. Πολύ ευχαριστώ θα απαντήσω στις ενδεχόμενες ερωτήσεις σας, όποτε επιθυμείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μορέλ. Είναι μεγάλη μου χαρά να καλωσορίσω την κυρία Αμονγκίν τώρα που είναι βουλευτής από την Ουγκάντα και βουλευτής του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, δηλαδή του ομολόγου μας στην Αφρική. Η κυρία Αμονγκίν θα μας μιλήσει για τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική ζωή στη χώρα της και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από πρώτο χέρι θα λέγαμε πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα της Έχετε το λόγο και εσείς για 10 λεπτά κυρία Μονγκίν. Χαίρομαι που ήρθατε. Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω όλους τους ε, συμμετέχοντες στο στρογγυλό τραπέζι, στο, στην, στην ακρόαση. Εγώ είμαι η Ζακλίνα Αμόγγιν και είμαι μέλος του Κοινοβουλίου στην Ουγγάντα και εκπροσωπώ την Ουγγάντα και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και ασχολούμαι με θέματα γεωργίας, φυσικούς πόρους, κουλτούρα και παιδεία και περιβάλλον. Ε, εγώ έγινα όταν ήμουν 24 ετών βουλευτής, ε, φρέσκια από το Πανεπιστήμιο έτσι απόκτησα πολλή εμπειρία σε ό,τι αφορά νομοθετικά θέματα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Στην Ουγκάντα και γενικά στην Αφρικανική Ήπειρο, όταν μιλάμε για συμμετοχή των νέων, πρέπει να πω ότι ε, κάναμε πολλά πράγματα για να προχωρήσει η σχετική ατζέντα. Υπάρχει πολιτική που διασφαλίζει τις ευάλωτες ομάδες. Ευάλωτοι τι, ποιοι είναι. Είναι αυτοί που δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν περιουσιακά στοιχεία, κάποια εχέγγυα. Οι νέοι, οι γυναίκες, οι άνθρωποι με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι επίσης. Αρχικά, όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια, παίξαμε ρόλο ως φοιτητές στην Αφρικανική Ένωση. Και δημιουργήσαμε, παίξαμε ρόλο για να δημιουργηθεί ο χάρτης για τους νέους στην Αφρική, που είναι το καθοδηγητικό έγγραφο που διέπει την δραστή των νέων στα κράτη-μέλη. Ε, εμείς έχουμε ε, ε, ε, οκτώ από όλα τα κράτη της Αφρικής που έχουν ε, επικυρώσει και χρησιμοποιούν το χάρτη σε όλες τις δραστηριότητες για τους νέους. Πολιτική συμμετοχή, ε, ε, επιρροή για την πολιτική για τους νέους στα κράτη-μέλη. Η Ουγγάντα έπαιξε ρόλο υποδείγματος εις ό,τι αφορά την ένταξη των νέων στην πολιτική. Πολιτική ανοιχτών θυρών ακολουθήθηκε. με βάση το Σύνταγμα οποιοδήποτε είναι άνω του, των 18 ετών μπορεί να διεκδικήσει πολιτικό αξίωμα. Έτσι έγινα κι εγώ από τους νεότερους βουλευτές, βγαίνοντα από το Πανεπιστήμιο αμέσως. Τα συστήματα μας είναι ανοιχτά. Μπορεί κανείς ε, να αναλάβει αξιώματα σε τοπικό επίπεδο, σε επαρχιακό, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, νωρίς. Και στην Ουγγάντα, για παράδειγμα, Παρόλο που στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έχουμε και ε, ε ηλικιωμένα ε, στελέχη, εγώ 24 ετών μπήκα και στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ως νέοι πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς εμάς. Ε, δεν είναι μόνο ηλικία, είναι και ε, ο μεγάλος αριθμός των νέων. Όλοι επηρεάζονται ε, από τις πολιτικές επιλογές. Στην ε, κοινότητα της Ανατολικής Αφρικής έχουμε και εκεί τον χάρτη των νέων που εξηγεί τη συμμετοχή των νέων. Δηλαδή 18 ε, και άνω στα διάφορα προγράμματα της κυβέρνησης και σε πολιτικούς τομείς ή ο Παναφρικανικός χάρτης, ο χάρτης της Ανατολικής Αφρικής ε, υπάρχει και στη Δυτική Αφρική ε, χάρτης και ε, όλα αυτά χρησιμοποιούν για να μετασχηματιστούν ε, οι βασικές αρχές της εθνικές πολιτικές. Είναι πολύ σημαντικό να εμπλέκονται οι νέοι στην πολιτική. Πώς θα γίνει αυτό με την ενημέρωση. Ε, ένας ενημερωμένος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί καλύτερα, μπορεί να αμφισβητήσει ε, γνωστές προσωπικότητες, ε, κυριάρχες πολιτικές. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τις θέσεις της κυβέρνησης, τον προγραμματισμό της, ε, ούτως ώστε να προωθήσει τα συμφέροντα της ε, ομάδας των νέων, την νεολαία της Αφρικής και της Ουγκάντα. Για να επηρεάσουν την πολιτική συμμετοχή οι νέοι στα κράτη-μέλη, πολλά μπορούν να γίνουν, όπως είπε η συνάδελφος Μορέλ. Υπάρχουν πολλά προγράμματα για νέους ανθρώπους και εταιρικέ σχέσεις Ένωσης Αφρικής. Είναι αρκετά έξυπνα αυτά τα προγράμματα και μπορούν να προσελκύσουν περισσότερους νέους για να συμμετάσχουν και να ενημερωθούν, για να παίρνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να επηρεάσουν την πολιτική διάσταση των κρατών μελών ή κάποιου συγκεκριμένου κράτους μέλους. Στην Ουγκάντα ε, είμαστε στο Κοινοβούλιο εδώ και 8 χρόνια και επηρεάσαμε τον πολιτικό προσανατολισμό εις ό,τι αφορά τους νέους Παλιά δεν υπήρχαν νέοι στους εκπρόσωποι στους διάφορους τομείς. Τώρα τα καταφέραμε. Πολλοί έχουν εκλεγεί άμεσα στο κοινοβούλιο. Ε, εγώ ε, έδωσα ε, προεκλογικό αγώνα για να εκλεγώ και υπάρχει πρόνοια για να προωθούνται νέοι. Και στα, στους ΟΤΑ ε, έχουμε άμεσα εκλεγμένους νέους ανθρώπους. Όταν είναι κανείς στο, στην κουζίνα μπορεί να αποφασίσει τι θα φάει. Όταν είναι στο σαλόνι δεν μπορεί, δεν έχει πρόσβαση. Κάτι τέτοιο θέλω να πω. Να βάλουμε στην κουζίνα νέους ανθρώπους, περισσότερους. Η Αφρικανική Ένωση μιλάει για την Ατζέντα 2063 αυτή θα επηρεάσει ακόμη περισσότερους νέους. Ο οι παππούδες μου ε, που πέθαναν όταν ήμουν τριών ετών ε, ε, δεν πρόλαβα να δουν αυτά. Σήμερα ζούμε περισσότερα. η συμπερίληψη των νέων που θα συμπεριλαμβάνουν στην κυβέρνηση, την πολιτική συμμετοχή είναι πολύ σημαντικό και εντάσσει τους νέους ε, σε όλους τους τομείς. Ε, στην περίοδο πριν από το Αμπιτζάν που θα δούμε τη σχέση Ένωσης Αφρικής ε, είναι σημαντικό να δούμε αυτό αν θέλετε το μέρισμα που προσδίδουν οι νέους. Η Ουγγάντα τώρα ε, έχει υιοθετήσει σχετικές πολιτικές για τους νέους. Στο τομεακό πρόγραμμα ε, που ετοιμάζομαι πριν ε, πάμε στο Αμπιτζάν θα μιλήσουμε και για την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το τομέα εντάσσομαι νέους στην πολιτική. Αν πιάσουμε το θέμα της και αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή περιορίζεται και η μετανάστευση, γιατί υπάρχει και κλιματική μετανάστευση λόγω αλλαγή του κλίματο, Φεύγει ο κόσμο και εγκαταλείπει τι αιστείε του. Θα ήθελα να σα πω ότι στην Ουγγάντα το 70% είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 45 ετών. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε αρνητικό για την οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή τους, οτιδήποτε αρνητικό πλήττει περισσότερο τους νέους. Γι' αυτό τα θέματα κλιματικής ε, αλλαγής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, εγώ έχω ένα, ε, δημιούργησα ένα ίδρυμα που φέρει και το όνομά μου στην Ουγκάντα και ασχολείται με παιδιά, νέες κοπέλες που φεύγουν πρόωρα από το σχολείο. Ένας άντρας μπορεί να συνεχίσει πιο εύκολα τις σπουδές, ενώ το παιδί θα παντρευτεί, το κορίτσι θα παντρευτεί, θα εγκαταλείψει τις σπουδές και κανέναν δεν τον πειράζει. Ενώ εμείς λέμε όχι, όλοι έχουμε δικαιώματα. Όλοι γεννηθήκαμε με τα ίδια δικαιώματα. Και στην παιδεία, παιδεία για όλους. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες, ε, τέτοιοι βιώσιμοι στόχοι. Υγεία, υγεία για όλους. Και υπηρεσίες που βοηθούν τις γυναίκες σε αναπαραγωγική ε, ηλικία. Ε, δεν πρέπει να προωθούνται περισσότερο τα άρενα από τα θύλαια ε, παιδιά. Θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση σε όλα αυτά. Με αυτές τις παρατηρήσεις σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο και χαίρομαι πολύ και για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα προχωρούμε στον τελευταίο μιλητή μας του, του, πρώτου γύρου και χαίρομαι που μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Μουνί Όρο που είναι συντονιστής προγράμματος της Εθνικής Ένωσης Οργανώσεων Νέων. Θα μας μιλήσει για τη, τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής Αφρικής Ένωσης για τους νέους. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα, οπότε ας ξεκινήσω λέγοντας το διεθνές πλαίσιο στις σχέσεις μας εξελίσσεται συνεχώς και το οποίο προσέζει ευκαιρίες και προκλήσεις από την πρώτη ασκήψη κορυφή στο Κάιρο το 2000 όπου το πλαίσιο εταιρικής σχέσης θεσπίστηκε έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές και στις δύο υπήρους που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η μία νεολαία αντιλαμβάνεται την άλλη. Θεσμοθετήθηκε λοιπόν η συνεργασία στον τομέα της νεολαίας μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρώτη ασκήψη που έγινε το 2007 για να αυξηθεί η συμμετοχή των νέων στην εταιρική αυτή σχέση. Σήμερα υπάρχουν πολύ περισσότεροι νέοι από ό,τι παλαιότερα στον κόσμο, 1,8 δισεκατομμύρια, κάτι το οποίο αποτελεί ένα άνευ προηγουμένου δυναμικό για οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Παραδόξως πάρα από τους, από αυτούς τους νέους ζουν σε ακραία φτώχεια, υψηλά, με ψηλά επίπεδα ανεργίας, περιορισμένη πρόσβαση στους πόρους, μισολοδοξία, έλλειψη συμμετοχή στη δικασία λήψη αποφάσεων, σειράξει κλπ. Η νεολαία λοιπόν στην Αφρική και στην Ευρώπη θα αντιμετωπίζουν αυτό ως καθημερινότητα καμιά φορά. Και μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση μέσω παροχής ευκαιριών και κοινοτομίας. Και αυτό ήταν και το θέμα επένδυση δηλαδή στην ΟΕΝΕΑ, στο τέταρτο στην τέταρτη σκέψη κορυφής Ευρω... Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είχαμε δημιουργία ενό διαλόγου, μιας πλατφόρμα διαλόγου όπου συμμετείχαν νέοι, οργανώσει νέων και οι πολιτικοί από την Ένωση και την Αφρική για να αντιμετωπιστούν οι κοινέ προκλήσεις. Να τονίσω ότι η επένδυση στην νεολαία αποτελεί μια προπόθεση για την οικοδομήση ενό βιώσιμου μέλλοντο στις διασυνδεδεμένες κοινωνίες μας. Χρειάζεται βεβαίως και στήριξη και όθηση της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και πρόσβαση της αγοράς. Η επένδυση στους νέους σημαίνει ότι θα πρέπει να παράσχουμε το σωστό πλαίσιο στους νέους ώστε να πετύχουν τις ε, φιλοδοξίες τους και να ελοποιήσουν τις δυνατότητε τους. Θα πρέπει επίσης να, επενδύσουμε και να διευκολύνουμε τους πολλαπλούς ρόλους που μπορούν να παίξουν στην, στην κοινωνία συμπεριλαμβανομένων και των γεφυρών μεταξύ κράτους και ε, νέων. Ιδιαίτερα στην Αφρική όπου βρίσκονται στο περιθώριο συχνά οι νέοι και δεν έχουν φωνή επιρροής. Η πρόσφατη διάσκεψη κορυφής επέτρεψε στους νέους και από τις δύο υπηρούς να τονίσουν μέσω έξι ψηφισμάτων σημαντικά θέματα που αφορούν και τις δύο υπηρούς και που περιλαμβάνονται στην κοινή δήλωση για την νεολαία που μεταβάστηκε στους, αρχού, στους αρχούς κρατών. Αφορούν την εκπαίδευση, την ασφάλεια και την ε, ειρήνη, ε, διακυβέρνηση, περιβάλλον, επιχειρηματικότητα, πολιτισμός. Έχουμε μια πρωτοβουλία λοιπόν που εμπλέκει τους νέους και από την Ένωση αλλά και από την Αφρική για την υλοποίηση αυτή του θεματολογίου. Στο Αμπιτζάν είχαμε προτάσεις για πρακτικές λύσεις και προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν μετά την διάσκεψη στο Αμπιτζάν. Και στην δήλωση Κάλεσαν οι νέοι του αρχηγού καρτών κυβερνήσεων τη Αφρική και τη Ένωση να καταβάλουν προσπάθειε να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στην συμμετοχή των νέων στην αγορά και την πρόσβαση των νέων στα δικαιώματα. Οι συστάσει τονίζουν την ανάγκη για την παροχή του σωστού περιβάλλοντο στου νέου, ώστε να υλοποιήσουν τι δυνατότητέ του και να έχουν αντίκτυπο στι κοινωνίε. Οι αφρικανικέ οργανώσει διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο εκπροσωπώντα την νεολαία τη που συχνά ε, είναι αντιμέτωποι με εκμετάλλευση, πολέμους και σοβαρές ασθένειες στην Αφρική. Για την ε, εκπαίδευση και τις δεξιότητες μίλησαν για την αναγνώριση των δεξιότητων τους που προέρχονται από την εκπαίδευση όπως επίσης και την γενική πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Θέματα που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές εδώ. Ζήτησαν λοιπόν οι συμμετέχοντες νέοι σε αυτές τις διασκέψεις να υπάρχει βιώσιμη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ώστε να δημιουργήσουν δυνατότητες capacity building. Η συμμετοχή επίση στην δημοκρατική διακυβέρνηση πρέπει να διέρχεται από τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητα σε εκλογές όπως ακριβώς στην Ευρώπη για να προχωρήσουν ακριβώς οι νέοι για να εξελιχθούν. Ζήτησαν λοιπόν οι εκπρόσωποι να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν και διακρίσεις στις δύο και τόνισαν τα κίνητρα τα οποία θα πρέπει να δοθούν στις ε, κοινοβουλευτικές ε, δημοκρατίες μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού η δήλωση ζητά από την εταιρική σχέση να προωθήσει την πολιτισμική παραγωγή προστατεύοντας και διατηρώντας όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες της ε, κοινωνίας αυτές. Επίσης, για την τέχνη και τον πολιτισμό να ενισχυθούν τα αφρικάνικα προγράμματα καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω επένδυσης, κατάρτισης, ε, προώθησης και παραγωγής ε, πολιτισμού για τους νέους. Να τονίσω ότι ο πολιτισμός αποτελεί το εργαλείο μεταβολής, μετατροπής ολόκληρων ε, κοινωνιών και αναζήτησης της ταυτότητας και του ανήκειν για όλες τις ηλικίε. Αποτελεί επίσης και ένα σοβαρό εργαλείο για την εμπλοκή των πολιτών. Δηλαδή ο πολιτισμός διδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και εργαλείο για την εξέλιξη των μελλοντικών κοινωνιών αποτελεί και ένα κύριο στοιχείο για την πρόθεση τη αμοιβαία πολιτικής κατανόηση και τη ειρήνης. Ε, σε αυτά θα πρέπει να φαίνεται λοιπόν η εταιρική μα σχέση και θα πρέπει να αποτελεί μια προπόθεση. Η επένδυση στου ε, τοπικού τοπικούς πολιτισμούς, τοπικέ τοπικές κουλτούρες και η χρήση πόρων για το θέατρο, τη μουσική, τα διάφορα φεστιβάλ μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών οικονομιών ώστε να δημορφωθεί σωστά η κοινωνική συνοχή και η ταυτότητα, τοπική ταυτότητα. Η πρόθεση της δημιουργικότητας μεταξύ των νέων είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα στην αναζήτηση λύσεων για τις σημερινές προκλήσεις. Συγγνώμη, ο μιλητής διορθώνω. Η δημιουργικότητα πέραν των άλλων πόρων αποτελεί ένα σημαντικό πόρο προώθησης κοινωνικής πρόοδους, πρόοδου για άτομα όλων των ηλικιών. Η θεσμικοποίηση αυτής της καλλιτεχνικής δημιουργίας βοηθά τους νέους να αντιμετωπίσουν τις κυριότερες προκλήσεις των κοινωνιών τους και βοηθά τους πολιτισμούς τους. Η Αραβική Άνοιξη μας έδωσε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία και τα διδάγματα μας έδειξαν ότι η δημιουργικότητα μπορεί να πάει στην επιχειρηματικότητα και στην κοινωνική συνοχή. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να έχουμε κοινωνική αστάθεια σε αυτές τις χώρες. Σήμερα βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας ε, άλλου ενός ε, παγκόσμιου μετασχηματισμού. Έχουμε την ε, γενιά των νέων επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά, σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά ε, το περιβάλλον, την βιωσιμότητα και άλλες σημαντικές προκλήσεις. Ο ρόλος λοιπόν του Κοινοβουλίου θα πρέπει να είναι κρίσιμος για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα σε επίπεδο ηθινόντων. Η χάρτα είναι πολύ σημαντική για τους νέους και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο τους επόμενους μήνες και χρόνια για θέματα που αφορούν προγράμματα για τους νέους. Είναι απαραίτητο να έχουμε συμφωνίες οι οποίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των νέων ώστε όλα αυτά να τους καταστήσουν αμοιβώς υποφελούς συνεταίρους και συνεργάτες ώστε να προχωρήσει και η δημοκρατία στην Αφρική υπέρ των πολιτών της, ιδιαίτερα υπέρ των νέων πολιτών της. Έχουμε λοιπόν ωφέλη τα οποία δεν μπορούν να αποκομιστούν μεμονωμένα χωριστά στην απομόνωση. Να παραθέσω και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Μπανκιμούν, ο οποίος έλεγε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ το δυναμικό που παρουσιάζει το 1,8 δις νέων παγκοσμίως αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να δώσουμε νέα φωνή, νέο ρόλο στο νέο θεματολόγιο και ένα κύριο σημαντικό ε, κυρία σημαντική συμμετοχή που θα μπορούσαν να έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές του πρώτου γύρου. Έχουμε τώρα περίπου 10 λεπτά για να μπορέσουμε να θέσουμε ερωτήσεις Δέκα λεπτά μάλλον για τις ερωτήσεις και μετά θα απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Και ας αρχίσουμε με την κυρία Φερχάιεν. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Ανακύπτουν αρκετά ερωτήματα. Πρώτα, τι γίνεται με την πρόσβαση στην εκπαίδευση και για νέα παιδιά από ευάλωτες ομάδες, από κοινότητες της υπαίθρου πώς καλύπτονται, πώς εξασφαλίζονται επαρκείς δομές για την παιδεία σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο και σε ορισμένες χώρες, ιδίως όπου σημειώνονται ελλείψεις στην παιδεία. Γιατί για μένα έχει μεγάλη σημασία οι νέες και οι νέοι να έχουν, να αποκτήσουν προσόντα μέσω της παιδείας, να μπορούν δηλαδή να σφυριλατήσουν τις ε, δυνατότητες που θα μπορέσουν να έχουν μετά για να βασιστούν στην υπόλοιπη ζωή τους, διότι και οι δύο πλευρές είναι σημαντικές. Να δοθεί χώρος στους νέους, να μπορέσουν να εισέλθουν στην πολιτική, να παίξουν τον ρόλο τους ε, στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων. Χρειάζεται όμως και το υπόβαθρο και την εκπαίδευση για να τα κάνουν αυτά με αίσθημα ευθύνη. Για μένα το βασικό ερώτημα είναι, έχει κάθε παιδί την δυνατότητα να πάει στο σχολείο να απολαύσει την εκπαίδευση, να μπορέσει να αναπτύξει τα ταλέντα του. Ποια είναι η κατάσταση για την ώρα. Σας ευχαριστώ. Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ. Αυτό που μας δώσατε σήμερα είναι μια πολύ θετική όψη των νέων και των γυναικών από την Αφρική μια κινητήρια δύναμη θαυμάσια αλλαγή και σας ευχαριστώ για αυτές τις θαυμάσιες μαρτυρίες σας. Ευχαριστώ και την κυρία Μορέλ για την ξεκάθαρη της αρχική τοποθέτηση. Έχουμε ερωτήσει και έχουμε και κάποιες επαληθεύσει που θέλουμε να κάνουμε μαζί για αυτές τις μεγάλες ευκαιρίε. Υπόθηκε ότι σε πολλέ αφρικανικές χώρες, 29, δόθηκε προτεραιότητα στην εκπαίδευση και έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Υπάρχουν όμως κάποια κενά όσον αφορά τα κορίτσια και τη δυνατότητα μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατάρτιση των εκπαιδευτών έχω διαβάσει κάποια πράγματα. Είναι λοιπόν σημαντικό εμείς εδώ να κάνουμε μια παλήθευση, μια αξιολόγηση των δύο προγραμμάτων και θα ήθελα εδώ τις απαντήσεις σας. Το Erasmus Mundus που πρασπίστηκε το κοινοβούλιο έστω και τα στοιχεία είναι περιορισμένα και το κομμάτι που αφορά τις νέ, τρεις νέες προτεραιότητες. Αυτό που υπόθηκε από εσά νομίζω ότι είναι καρπός συνεργασίας αυτό που έχουμε σε επίπεδο πολιτισμού και αυτό το είπε και ο κύριος Μουνιόρο προηγουμένως έχουμε διεθνή συνεργασία που προβλέπει τρία πράγματα για την κινητικότητα. Καταρχάς, ένα νέο πρόγραμμα κινητικότητας των νέων καλλιτεχνών, νέων δημιουργών, νέων φορέων του πολιτισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην διάσκεψη Ευρώπης, Αφρικής στο Αμπιτζάν θα μπορούσε να έχει κάποιους καρπούς και θα ήταν καλό να ακούσουμε και κάτι παραπάνω από την Κομισιόν γι' αυτό. Ένα άλλο σημείο αφορά τους νέους που σήμερα πρέπει όντω να ενταχθούν στις διαδικασίες πολιτικής εκπροσώπησης. Ξέρω ότι υπάρχει διαφορά στην ηλικία όσον αφορά το να είναι ερετή, να είναι υποψήφιοι αυτό ήθελα να ρωτήσω επίση, να πείτε τι γίνεται με αυτή τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ως μέλος της Επιτροπής ε, και ως συντονιστής της ομάδας μου, τα θέματα της ανάπτυξης ε, με απασχολούν ε, ιδιαίτερα στα πλαίσια της νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Ε, σε όλα αυτά τα προγράμματα οι νέοι είναι στο επίκεντρο και η πρόσβαση στην παιδεία πολύ σημαντική. 60% των 60% ε, του πληθυσμού της Αφρικής είναι κάτω από 25 χρονών. Και έτσι δημιουργείται ένα τεράστιο εργατικό δυναμικό που θα ασκήσει πιέσεις. Έτσι η εκπαίδευση και η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Ε, σημαντική επίσης είναι η επιμόρφωση. πέρα από τη, ε, ε, ε, όταν μιλάμε για την κατάσταση στο, των νέων στην Αφρική πρέπει να μιλήσουμε και για την εσωτερική μετακίνηση. Ε, θα αυξάνονται περισσότερο στο μέλλον και πολλοί δηλαδή μένουν στους προσφυγικούς καταβλισμούς. Τώρα, η πρωτοβουλία ε, στο Αμπιτζάν, η Αφρικανική Ένωση ε, έκανε ε, προτάσεις σχετικά με την κινητικότητα, την δυνατότητα εκμάθησης ε, επαγγελμάτων. Εμείς μιλάμε για τους βιώσιμους αναπτυξιακούς στόχους ο πέμπτος στόχος αναφέρεται στην ισότητα των φύλων. που είναι ένας βασικός νομικός κανόνας Στην Αφρική έχουμε ε, συχνά φαινόμενα ε, αναγκαστικών ε, γάμων, αμβλώσεων κλπ. Ε, σίγουρα είναι ένα θέμα κουλτούρας, αλλά ε, αυτά, τα θέμα, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την εκπαίδευση. Η κυρία Σιόρντοβα, ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι οι επενδύσεις ε, στους νέους είναι επενδύσεις στο μέλλον. η επένδυση στους νέους στην Αφρική είναι σημαντική και για μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση στην κυρία Μορέλ. Η ειρήνη νομίζω είναι η προϋπόθεση για όλες τις άλλες προτεραιότητες. Αλλά χωρίς ε, μορφωμένους νέους στην Αφρική δεν μπορούμε να χτίσουμε σε άλλες προτεραιότητες από αυτές που είπατε. Τι προϋπολογισμό έχουν αυτές οι προτεραιότητες αυτές, δηλαδή προχωρημένη γνώση και δεξιότητες. Ε, είναι ένα, τι ποσοστό είναι στα πλαίσια του Erasmus Συν, αν έχετε στοιχεία. Και μία ερώτηση στην κυρία Μοντζίν. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε ε, ένα κομμάτι από την πείρα σας ως πολιτικού. Ε, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις που θα βελτιώσουν τη συνεργασία και τη θέση των νέων στην Αφρική και στον κύριο Μουνιόρο Εσείς εργάζεστε με οργανώσεις νέων. Ποιος είναι ο βασικός σας εταίρος, ας πούμε, αν έχετε κάποιους εταίρους. Ε, με προσκόπους έχετε εμπειρία Ευχαριστώ. Η Watts, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Ήμουν και στο χθεσινό πάνελ για τη μετανάστευση. Ε, Ζακλίν, πραγματικά είστε πηγή έμπνευση. Χάρηκα πολύ που είχα την ευκαιρία να σας ακούσω. Ήταν προνόμιο. Έχετε να διδάξετε πολλά στους νέους στις ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί νέοι τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματά τους τα θεωρούν δεδομένα και δεν παλεύουν για αυτά. Και εν πολλής, ε, και εμείς δεν ε, τους κάνουμε σωστή αγωγή πολίτου ώστε να καταλάβουν ότι μπορούν να είναι μέρος της πολιτικής διαδικασίας. Εσείς είστε ένα λαμπρό παράδειγμα. Ε, στη χώρα σας ε, ποια είναι η κατάσταση ε, σε ό,τι αφορά τις οργανώσεις που ενισχύουν την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις που προσπαθούν να προωθήσουν και να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχα πάει στην Κένια για να παρακολουθήσω τις εκλογές ε, στα πλαίσια μιας αποστολής Φαίνεται να είναι σταθερή η χώρα, αλλά ήταν, αλλά τώρα ε, έχει εκτραπεί στη βία. Αυτή η βία μαθαίνω ότι προϋπήρχε, αλλά ήταν κρυμμένη από τα ΜΜΕ. Επίσης, ως καλλιτέχνης ε, η ίδια, πιστεύω ότι οι τέχνες και ο αθλητισμός, ε, ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις, τη βία, να ε, προχωρήσουμε στην ειρήνευση. Καλό είναι να δούμε προληπτικά και εκεί μπορεί να βοηθήσει ο πολιτισμός και οι τέχνες και η συνεργασία με τους νέους των διαφόρων κοινοτήτων. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε τη σύγκρουση αντί να μαζεύουμε μετά τα κομμάτια της σύγκρουσης. Ευχαριστώ ο κύριος Νεκόφ. Ε, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά τις ε, τοποθετήσεις σας. Μιλήσατε για τους νέους, για την ανάπτυξη, για τις συγκρούσεις. Χθες μία νέα μας είπε ότι η πολιτική για την νεότητα δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός. Οι νέοι δεν είναι μονάχα πρόσωπα που πρέπει να εκπαιδευτούν, δεν είναι μόνο το μέλλον. Οι νέοι και οι νέες είναι και η δυνατότητα που έχουμε να διατηρήσουμε την ειρήνη οι άνθρωποι που θα αναλάβουν την επιστημονική έρευνα. Αλλά οι ναι, νέοι έχουν μια διαφορετική εικόνα του κόσμου. Κάποτε λίγα χιλιόμετρα ήταν ε, ανυπέρβλητο εμπόδιο απόσταση δηλαδή. Τώρα διανύουμε εκατοντάδες χιλιόμετρα σε ελάχιστο χρόνο η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής θα πρέπει να βασιστεί σε άλλες παραμέτρους. Οι πόροι, η χρήση των πόρων θα πρέπει να είναι στοχευμένοι. Οι χρήση των πόρων, οι χρηματοδοτήσεις δεν μπορούν να παραδίδονται απλώς στα χέρια των αφρικανικών κυβερνήσεων, θα πρέπει να κατευθύνονται σε ενώσεις, σε ομάδες που θα επιτρέψουν την δημιουργία νεοφιών επιχειρήσεων, start-up, την ε, δημιουργία συγκεκριμένων έργων. Άρα τα χρήματα να μην παραδίδονται ανεφόρων στα χέρια των ε, κυβερνήσεων, αλλά ξαναλέω να στοχεύουν στην διευκόλυνση κοινών πρωτοβουλειών που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της Αφρικής. Ένας νέος Σουδανός, νεαρός δηλαδή, ε, εργάζεται στην Βουλγαρία και έχει δημιουργήσει μια επιχείρηση που παράγει προϊόντα τα οποία επανεξάγονται στην Αφρική. Υπάρχουν πολλά επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία μπορεί κανείς να ε, ε, χρησιμοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νεκόφ. Δεν θέλω να σας κόψω το λόγο λόγω αυστηρότητας, αλλά είναι λίγο δύσκολο να τηρήσουμε τα χρονικά μα πλαίσια. Και γι' αυτό τώρα θα είναι και λίγο δύσκολο το καθήκον των τριών πρώτων εμπειρογνωμόνων μα να απαντήσουν στι πολλέ παρατηρήσει σα. Αλλά δεν είστε και υποχρεωμένοι να, να απαντήσετε σε όλε. Μπορείτε να επιλέξετε εκεί όπου θεωρείτε ότι μπορείτε να συμβάλλετε καλύτερα στην αύξηση των γνώσεών μα. Θα έλεγα λοιπόν να αρχίσουμε από την, με την αντίθετη σειρά και να αρχίσουμε επομένω με τον κύριο Μουνιέρο. Μουνιόρο, συγγνώμη. Δύο λεπτά, κύριε. Σας ευχαριστώ να απαντήσω στο τελευταίο θέμα που είπατε για την συμμετοχή των νέων στην ανάπτυξη. Όπως λέει και η διακήρυξη, οι νέοι στηρίζουν την ε, διακήρυξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια και ειρήνη και ασκούν και πίεση προς την κατεύθυνση αυτή. Ρωτήσατε και για τη δουλειά που κάνουμε και για τους σημαντικότερους εταίρους μας που μας βοηθούν. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε τοπικό γραφείο στην Ζιμπάμπουε, έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας επιτρέπει να συνεργαζόμαστε για θέματα ανάπτυξης, δημιουργίας ε, των συνθήκων για την ειρήνη, για την εμπλοκή των νέων και ένα θέμα το οποίο τέθηκε για την συμμετοχή των νέων στην πολιτική. Στην χώρα όπου, από όπου κατάγομαι, οι νέοι είναι το 67,7% του πληθυσμού. Συχνά είναι όμως απαθείς, είναι απογοητευμένοι σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στα κοινά. Και αυτή μάλιστα είναι και η γενικευμένη εικόνα στην Αφρικανική Ήπειρο. Δηλαδή δεν ε, καταλαμβάνουν τον χώρο που θα έπρεπε σε θέματα της κοινωνίας οι, οι νέοι. Τελευταία μου απάντηση σχετικά με την πρόσβαση των νέων και ιδίως από τις περιοχές της Υπέθρου στην παιδεία. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχουμε περισσότερα κορίτσια. Όσο προχωρεί κανεί όμω προ τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σιγά σιγά προ τα πανεπιστήμια, βλέπουμε όλο και περισσότερα κορίτσια να εγκαταλείπουν. Και εν τέλει βλέπουμε μία τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Ε, και αυτό οφείλεται σε κάποιε δομικέ διαφορέ. Ευχαριστώ η κυρία Αμονγκίν. Δύο λεπτά, κυρία Αμονγκίν. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας. Και θα απαντήσω στην ερώτηση για την πρόσβαση στην ε, παιδεία και το θέμα του φίλου Στις περισσότερες χώρες το αρσενικό φύλο παίζει σημαντικό ρόλο ακόμα στην, ε, και στην παιδεία όπως και γενικότερα στην κοινωνία όταν φτάσετε στην ηλικία των 18 στις περισσότερες κοινότητες, ακόμη και στην Ουγκάντα, αναμένει η κοινωνία το κορίτσι να παντρευτεί, το αγόρι να συνεχίσει. Το κορίτσι θα μείνει στην κουζίνα να μαγειρεύει. Στο χωριό μου ήμουν η πρώτη απόφυτος και όταν έλαβα το πρώτο μου πτυχίο, πτυχίο ε, αισθανόμουν άσχημα διότι τα άλλα κορίτσια, οι συμμαθήτριές μου, είχαν ήδη 7 παιδιά και ήμασταν μόνο 19 χρονών. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι κοινότητες αυτές την ανάγκη να προχωρήσουν και τα κορίτσια και τα αγόρια στο σχολείο. Να αλλάξει απλώς η αντιμετώπιση που έχει η κοινωνία. Διότι το πατριαρχικό μοντέλο παίζει ακόμα πολύ σημαντικό ρόλο. Και όταν πήγα στο κοινοβούλιο μας το πρώτο νομοσχέδιο που κατέθεσα η πρώτη πρόταση νόμου δηλαδή ήταν αγόρια και κορίτσια να παίξουν ισότιμο ρόλο στην παιδεία. Αυτό τώρα έχει υλοποιηθεί, όμως η διαδικασία είναι σταδιακή, δεν έχουμε πάει πολύ μακριά. Πρόκειται για συλλογική προσπάθεια και μια και μιλούμε και για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απαραίτητο να γίνει το mainstreaming των φύλων. Άλλο είναι ότι 29 χώρες της Αφρικής έχουν αναλάβει δέσμευση για την παιδεία. Όμως και οι 54 αφρικανικές χώρες έχουν συνυπογράψει τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμεύονται. Όμως, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών και το πλαίσιο στο οποίο έχουμε ενταχθεί, οι προσδοκίες ακόμα είναι πολύ χαμηλές. Να περάσουμε από τα λόγια στην δράση εφόσον έχετε δεσμευτεί, μπορείτε να δεσμευτείτε και ότι θα αποδώσετε την αναγκαία προτεραιότητα. Ε, <laughs> με συγχωρείτε, λέει η κυρία Μονικινά, μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ωραία. Ε, πρόκειται για ένα χώρο που ε, υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούμε κι άλλο. Επίσης, το θέμα του γάμου των νέων κορισιών και αν θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους του 2063 θα, ε, αν δεν πάνε όλα τα παιδιά στο σχολείο δεν θα έχουμε τα αναγκαία βασικά αγαθά και δεν θα ε, ολοκληρωθούν οι στόχοι της Ατζέντα 2063. Να με συμπαθάτε που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα απλώς να σα επιτρέψω να δειτε ολόκληρο την πρότασή σας, μην αρχίσετε όμως κι άλλοι. Ε, τώρα, η κυρία Μορέλ, δύο λεπτά σας παρακαλώ κυρία Μορέλ, να απαντήσω συγκεκριμένα σε μια ερώτηση για τον προϋπολογισμό που αφιερώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ε, παιδείας, εκπαίδευσης, πρόσβασης αναφερόταν και σε μια από τις διαφάνειες ήταν 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ για την παρούσα προγραμματική περίοδο και εκτός από αυτού και, και, και, αυτό μάλλον ε, δίνεται για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών πρόσβαση στην παιδεία επαγγελματική και ε, εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαίδευση των εκπαιδευτικών των δασκάλων δηλαδή γιατί αν δεν αρχίσετε να ενισχύσετε την ε, εκπαίδευση των δασκάλων δεν ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά ο στόχος όπως είπα 1,34 δισεκατομμύρια ευρώ και εκτός αυτών είναι και τα χρήματα που δίνονται στο πρόγραμμα Erasmus και αυτό κατευθύνεται και στις χώρες υποσαχάριας Αφρικής και για τον Erasmus δίνουμε εκεί 300 εκατομμύρια και ο Erasmus στο στοχεύει κυρίως στην ανώτερη εκπαίδευση και στην άτυπη εκπαίδευση και όλες τις μορφές της άτυπης μάθησης. Και όπως είπα, αυτό είναι τμήμα αυτής της συνολικής προσέγγισης. Δηλαδή δεν εξετάζουμε μονάχα την τυπική εκπαίδευση που γίνεται μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Μιλούμε ακόμη για την ε, εκπαίδευση στο επιχειρήν ε, ε, γυναικών και νεαρών κοριτσιών πώς να αντιμετωπίσουν δηλαδή τις επιχειρηματικές τους ικανότητες και όχι μόνο ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς πληθυσμούς αλλά και στις τοπικές κοινότητες. Και πάλι μιλώ για εκπαίδευση των δασκάλων, συνεργαζόμαστε με τα πανεπιστήμια εκεί και χρειαζόμαστε βεβαίως γιατί πολλοί από τους δασκάλους εκπαιδεύονται σε αυτά τα πανεπιστήμια και πρέπει να διατηρηθεί η επαφή με τους τοπικούς πληθυσμούς. Πρέπει να δούμε πώς θα διευκολύνουμε την πρόσβαση αυτή. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία όχι μόνο με τα εθνικά υπουργεία και άλλες εθνικές αρχές, αλλά πρέπει να φτάσουμε μέχρι το επίπεδο των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών αρχών και στην Ήπεθρο, όπου το ζήτημα της πρόσβασης είναι βέβαια ιδιαίτερα κρίσιμο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της ανταλλαγής απόψεων και αρχίζομαι με ένα πολύ σημαντικό θέμα, δηλαδή εκπαίδευση και αθλητισμός, η περίπτωση της Νιγερίας. Ο κύριος Λά είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής της ε, Γερουσίας για την άμβληση της φτώχειας και την κοινωνική πρόνοια. Ε, έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδρε της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Επαιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Κάμερεφερτ. Διακεκριμένη Διακεκριμένοι συνάδελφε από το Κοινοβούλιο της Ουγγάντα, κυρία Μογκίν. Χαιρετίζω επίσης τον αναπληρωτή διευθυντή, Γενικό Διευθυντή για την Αφρική, της UNESCO, ε, αγαπησιότιμα μέλη, μέλη του διπλωματικού σώματος. Είναι μεγάλη χαρά που έχω προσκληθεί σε αυτό το πρόγραμμα και έχω τη δυνατότητα να εκφράσω τις σκέψεις μου σε ένα σημαντικό θέμα. Το θέμα της παιδείας και του αθλητισμού στις δύο υπήρους μας, που τώρα έχει αποκτήσει περισσότερη σημασία από ποτέ. Η αναγνώριση των ωφελών της παιδείας και του αθλητισμού ε, μας επιτρέπει να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα προς ε, ένα κόσμο με περισσότερη φιλία και συνεργασία. Η Ευρώπη έχει καλύτερη κατανόηση του αθλητισμού και της παιδείας ίσως και έχει ωφεληθεί από αυτά πολύ περισσότερο από ότι η Αφρική. Οπότε δεν υπάρχει καλύτερος χώρος για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και ελπίζω να αντλήσουμε και κάποια θετικά διδάγματα και να έχουμε καλύτερη συνεργασία από ότι αυτό εδώ το βήμα. Γι' αυτό ελπίζω ότι θα συμμεριστώ κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις ελπίδες μας για να επιδιώξουμε θετικούς τρόπους να βελτιώσουμε τα θετικά της καλύτερης παιδείας. Γι' αυτό και έχω επιλέξει το θέμα παιδεία και αθλητισμός η περίπτωση της Νιγηρίας. Η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη κάθε κοινωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα που έχουν τα μέλη της κοινωνίας αυτής, ιδιαίτερα των νέων, να εκπαιδεύονται και να συμμετέχουν σε γόνιμη απασχόληση. Η εκπαίδευση και η απασχόληση διασφαλίζει ότι τα μέλη της κοινωνίας θα μπορούν να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινωνίας. Η σημασία της ύπαρξη μιας κοινωνικά δίκαιης κοινωνίας όπου η καλή εκπαίδευση και η συμμετοχή στον αθλητισμό μπορεί να συμβάλλει είναι σημαντική και κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα της Νιγερίας. Ιδιαίτερα το κεφάλαιο 2 με τις κατευθυντήριες γραμμές και τους στόχους για την κοινωνική δικαιοσύνη. Ένα, μια διάταξη κλειδί σε αυτό το κεφάλαιο είναι η απέτηση για τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευση για όλους τους πολίτες και η δημιουργία περιβάλλοντος καλής υγείας. Το αθλητισμός είναι ενσωματωμένο στα αναλυτικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ιγερία λοιπόν. Ε, για παράδειγμα, η Εθνική Πολιτική για την Εκπαίδευση αναγνωρίζει την ανάγκη κάθε παιδί στην Ιγερία σε όλα τα επίπεδα της ε, εκπαίδευσης να συμμετέχει στον αθλητισμό. Και υπάρχει μεγάλη έμφαση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Ε, είναι η φυσική αγωγή και το μάθημα της υγιεινής είναι υποχρεωτικά στα γυμνάσια και προαιρετικά είναι μόνο στα λύκεια. Με άλλα λόγια, η νιγηριανή πολιτική παιδεία πάντα αναγνώριζε τη σημασία του αθλητισμού. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πολλές φορές δυσκολευόμαστε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Δεν έχω χρόνο να μιλήσω για την σχέση παιδείας και αθλητισμού στην Νιγηρία. Θα μιλήσω περισσότερο για την παιδεία, γιατί έτσι κι αλλιώς ε, είναι παρόμοιες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στους δύο τομείς και με παρόμοιο τρόπο επηρεάζουν και τους νέους. Σημαντικό είναι ότι η ανάπτυξη στην παιδεία θα οδηγήσει βελτίωση και στον αθλητισμό. Η παιδεία και η ανεργία στην Ιγυρία. Ένα σύμπτωμα κλειδί για την κακή παιδεία στην Ιγυρία είναι η ανεργία. Η ανεργία ως σύμπτωμα ελλειπούς αξιοποίησης των φυσικών και των ανθρωπίνων πόρων αναγνωρίζεται ως μεγάλο εμπόδιο ε, για την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση όλων των χωρών. Όλοι οι σχολιαστές για την ανεργία συμφωνούν ότι μια μείωση στο ποσοστό ανεργίας μπορεί ως επιτοπλίστων να επιτευχθεί μέσα από την παιδεία και αυτό με τη σειρά του θα δώσει έναυσμα για ανάπτυξη και πολιτική συμμετοχή. Στην Ιγυρία, όπως στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ανεργία κυρίως των νέων λόγω της κακής, ε, ε, των, των κακών ευκαιριών εκπαίδευσης. Αυτή η κακή εικόνα φαίνεται να ισχύει στις περισσότερες αφρικανικές χώρες και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό γιατί πρέπει να αναλάβουμε δράση. Οι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η ανεργία των νέων έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην κοινωνία. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι επιπτώσεις. Αύξηση στο ποσοστό εγκληματικότητας, ευαλωτότητα των ηλικιωμένων, γενική οικονομική στασιμότητα, συγκρούσεις, αρβεβαιότητα, ανασφάλεια, κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις στο Δέλτα του Νίγηρα και οι δραστηριότητες της Μπόκο Χαράμ στα βόρεια-ανατολικά συνδέονται με την ανεργία και την κακή εκπαίδευση. Ε, αυτοί οι νέοι που πλήττονται, που περισσότερο και επηρεάζονται, είναι άνεργοι, δεν είναι εκπαιδευμένοι και έτσι έχουν σύγχυση και αγανακτούν ενάντια στην κυβέρνηση. Ε, δεν είναι μόνο στην Ιγυρία αυτό. Για παράδειγμα, μια έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ανεργία των νέων δείχνει ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά μεταξύ των νέων αυξάνεται με την αύξηση της ανεργίας. Ε, αυτό δείχνει ε, και αυτό συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχει τόσες κοινωνικές υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, επειδή στην Ιγυρία οι νέοι δεν έχουν τέτοιες ευκαιρίες όπως έχουν οι νέοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι πιθανό να νιώθουν ακόμα πιο εγκαταλειμμένοι, αγανακτισμένοι και έτσι είναι επιρρεπεί στο έγκλημα. Περισσότερο από ότι η ομολογοί τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Ευρώπη. Πιθανόν ένα μακροπρόθεσμο ε, αποτέλεσμα του προβλήματος ε, είναι ότι η ανεργία των νέων μπορεί να οδηγήσει σε μικρή απασχόληση πριν από την συνταξιοδότηση και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις μεγάλες ηλικίες και έχουμε έτσι έναν ε, φαύλο κύκλο έλλειψης παιδείας, μία απασχολησιμότητας, εξάρτησης, φτώχειας, πολιτικής απάθειας και ροπή στο, στη βία. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων στην Ιγυρία. Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην συνεχιζόμενη αύξηση της ανεργίας στην Ιγυρία είναι πολλοί. Είναι συστημικοί παράγοντες, δηλαδή εμπόδια λόγω του στεγνού και μη προοδευτικού συστήματος παιδείας στην Ιγυρία. Στη, στον τομέα της κατάρτισης έχουμε ε, πολύ πτωχά εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα τα οποία δεν ετοιμάζουν τους νέους για την επιχειρηματικότητα και αυτό είναι μια ηρωνία γιατί και οι εργοδότες ε, τροφοδοτούν αυτή την κατάσταση, έχουν μια προκατάληψη εναντίον των επαγγελματικών εκπαιδευτικών τίτλων και προτιμούν την ε, ε, τις πρακτικές δεξιότητες. Ε, πολλές φορές απαιτούν πείρα ακόμα και από κάποιον που για πρώτη φορά πιάνει δουλειά. Έτσι, οι καινούργοι πτυχιούχοι δεν μπορούν εύκολα να βρουν αμοιβόμενη απασχόληση γιατί η απασχόληση ανακυκλώνεται ανάμεσα στους εργοδότες και η μάζα των ανέργων αυξάνεται. υπάρχουν και διαρθρωτικοί παράγοντες. Ε, οι πολιτικοί δεν ε, αντιλαμβάνονται τη σημασία της εκπαίδευσης και των άτυπων ε, τομέων. Για παράδειγμα, 54% ε, των θέσεων εργασίας στην Ιγυρία δημιουργούνται από τους άτυπους τομείς. Και είναι και αυτό ηρωνικό, μια ηρωνία, ένα παράδοξο, γιατί είναι περίπου, είναι ως επιτοπλίστων η ε, τομείς που δεν προωθεί η πολιτική παιδείας. Ε, ε, έχουμε πολλούς νέους που θέλουν να γίνουν συγκολητές ή να έχουν κάποια βιοτεχνικά επαγγέλματα αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν καλύτερα γιατί υπάρχει μια προκατάληψη ότι όλοι θα πρέπει να βρουν ανώτερα επαγγέλματα στις τράπεζες και στις ε, πετρελαϊκές εταιρείες. Αυτό υπάρχουν και περιορισμοί στις υποδομές. Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό για την ανεργία. Μία Η κακή εκπαίδευση σε συνδυασμό με τα προβλήματα υποδομών ε, αυξάνει την ανεργία. Δηλαδή ε, δεν υπάρχουν ε, ευρωπα... βιομηχανικές ζώνες, δεν υπάρχει υδροδότηση δικτύου, ηλεκτροδότηση και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Πολλοί ε, προτείνουν κάποιες προσεγγίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργική εκπαίδευση ε, και θα μειώσουν την ανεργία στην Ιγυρία, όπως η υποχρεωτική μαθητεία. Η Νιγεριανή κυβέρνηση έχει ήδη προγράμματα όπως το N-Power και ο βασικός στόχος εκεί είναι η παροχή κατάρτισης στους ανέργους πτυχιούχους και μη πτυχιούχους. Ο βασικό στόχος είναι να μπορέσουν αυτοί που μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι στο τέλος ή να ε, προσλαμβάνουν εργαζομένους. Ε, εμείς ε, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτές τις πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να αρχίσουμε παρόμοια προγράμματα μαθητείας όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε οικοδόμηση ικανοτήτων, ε, αλλά ε, εδώ χρειάζεται και η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματοδότηση και ενίσχυση των δημοκρατικών μας θεσμών. Η Νιγηρία έχει πολλά αναξιοποιητά ταλέντα, κυρίως στα πανεπιστήμια, σε όλους τους τομείς φυσικές επιστήμες, τη γεωργία, κοινωνικές επιστήμες και εδώ η Ευρώπη μπορεί να μας βοηθήσει να, ανοίξουμε τις, ε, ε, να ανοίξει αγορές για τα προϊόντα μας. Ε, αυτό θα βοηθήσει, θα αποτελέσει ένα κίνητρο για την καινοτομία, διότι βεβαίως όλοι θα ελπίζουν ότι θα έχουν αυξημένη κερδοφορία και πρόσβαση σε ανταγωνιστικές αγορές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η Σελίν Φαμπρικέτ, η οποία είναι Γενική Διευθύντρια του Δικτύου Νέων Επαγγελματιών χωρώνα και Ευχαριστώ που ήρθατε. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας και ευχαριστώ που δώσατε την ευκαιρία για τιμή να μιλήσω για αυτά τα θέματα εν ώψη και της διάσκεψης του Αμπιτζάν. Μη γραμματέας λοιπόν στο δίκτυο αυτό της Ευρωπαϊκής συγγνώμη, της ε, πλατφόρμας που επιτρέπει στους νέους να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες και να απολαύσουν ευκαιριών για την ένταξή τους στις παραγωγικές διαδικασίες. Συμμετέχουμε συμβουλευτικά σε άλλες πρωτοβουλίες και φόρουμ και συνεργαζόμαστε, συνεργαζόμαστε εδώ και καιρό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε την Αφρικανική Εβδομάδα που διοργανώνουμε με τους σοσιαλιστές. Έχουμε το Φόρουμ Νέων και συνοργανώνουμε την διάσκεψη νέων Πρέπει να σας πω ότι σήμερα με απογοητεύει κάπως η χαμηλή παρουσία βουλευτών. Παρ' όλα αυτά ελπίζω ότι η εισήγησή μου θα σε επιτρέψει να υποστηρίξετε τη δήλωση και να προωθήσετε τα θέματα που αφορούν τους νέους. Τον περασμένο Οκτώβρη είχαμε 120 εκπροσώπους των νέων που συμμετείχαν στην σύνταξη ισορροπημένων και εφικτών συστάσεων ώστε οι οργανώσεις νέων στην Αφρική και στην Ευρώπη αλλά και αλλού να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να αυξηθεί η επένδυση προς τις προς τις δραστηριότητες των νέων ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τη συμμετρική σχέση και συμμετοχή των νέων πώς να αντιμετωπίσουμε δηλαδή, την ανεργία των νέων και να τους επιτρέψουμε να συμμετάσχουν σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η, Ευρωπαϊκή, η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επικεφαλής ε, ε, χωρών και κρατών και κυβερνήσεων δεν θέλουν μόνο να ε, να έχουν επαφές αλλά και να κάνουν κάτι το συγκεκριμένο για το μέλλον των νέων όλων. Πρέπει να δούμε λοιπόν και τι γίνεται με τη συμμετοχή των νέων. Ερχόμενοι εδώ, θεωρώ ότι καταρχάς έχουμε ένα πρώτο βήμα για την υποστήριξη της συμμετοχή των νέων. Ας μην είμαστε όμως ε, αυτάρεσκοι. Θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, θα πρέπει να είμαστε ευρηματικοί, γιατί νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που αφορά τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα και τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει όμως έλλειψη αναγνώρισης τη προσθεμένη αξία και η τελική σχέση μεταξύ νεολαία της διασποράς της Αφρικανικής και της ε, Ευρωπαϊκής θα μας ε, επιτρέψει να περλάβουμε και άλλους, δηλαδή οργανώσεις, κυβερνήσεις, ώστε ό,τι κάνουμε να συνοδεύονται και από τα απαραίτητα κονδύλια. Τέλος, νομίζω ότι μια καλή εταιρική σχέση βασίζεται στην παρακολούθηση και στην συνέχιση της συνεργασίας. Τώρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μέσω εθνικών, περιφερειακών και άλλων καναλιών. Παρ' όλα αυτά, η αναγνώριση των νέων ως εταίροι είναι κάτι το οποίο προσφέρει σε αξία για το μέλλον και αυτό λείπει αυτή τη στιγμή. Έχουμε εκδηλώσεις για τους νέους κάθε δύο χρόνια. Έχουμε πάνω από 7.000 ε, νέους στην Ευρώπη και από την Διασπορά όπου συζητούν μέσω διαφορών εκδηλώσεων το πώς θα επιλύσουν διάφορα ε, ζητήματα της καθημερινότητας, της κρίσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιους ε, πρεσβευτές ανάμεσα σε αυτούς τους 7.500 ε, συμμετέχοντες για να συμμετάσχουν σε διάφορες εκδηλώσεις εδώ στο Κοινοβουλίο και συνεδριάσεις. Είχαμε και ένα πρόεδρο, ο οποίος ορίστηκε ως πρέσβης διαφορετικότητας. Παρόλα αυτά δεν έχουν υπάρξει συγκεκριμένε δράσει, δεν έχει υπάρξει πρωτοβουλία για την παρακολούθηση αυτών των πράξεων. Και τώρα, το 2018, έχουμε νέε δράσει. Θα πρέπει η Ένωση να θεωρήσει ότι αυτά τα θέματα έχουν σημασία. Δεν είναι απλά και μόνο θέμα παρακολούθησης και συνέχισης. Θα πρέπει να πούμε ότι συχνά μας λένε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια και δεν υπάρχει δυνατότητα διάχυσης των κονδυλίων λόγω περιορισμών. Ελπίζω λοιπόν ότι η επόμενη συνάντηση και η πρωτοβουλία που θα ακολουθήσει τις πρωτοβουλίες που έχουν προϋπάρξει να ευοδοθούν. Οι συστάσεις που είχαμε αφορούν ευρεία θέματα. Κυρίως όμως αφορούν τους στόχους που πρέπει να πετύχουμε. Γιατί και πάλι ξέρουμε ότι σε δύο χρόνια θα έχουμε άλλη μια διάσκεψη κορυφής νέων και θέλουμε αυτά τα πράγματα να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει χώρος για να περιλάβουμε ας πούμε την ψηφιοποίηση ως κύριο στοιχείο το οποίο θα προωθεί και θα επιτρέπει την εμπλοκή της ψηφιακής τέχνης στις αντιστοιχέ κοινωνίες. Το Ευρωπαϊκό μια ψηφιακή πλατφόρμα για την πολιστική ε, κληρονομιά βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για να εφαρμόσουμε την δήλωση, για να ολοποιήσουμε τη δήλωση του Αμπιτζάν. Νομίζω το θέμα εδώ δεν είναι να δημιουργήσουμε κάτι νέο, αλλά να βελτιώσουμε κάτι που προϋπάρχει. Η ευρωπαϊκή και η αφρικανική κουλτούρα είναι πλούσιες, όμως χωρίς αμοιβή αναγνώριση, χωρίς πρόθεση, χωρίς επένδυσης θα χαθούν αυτές οι κοινέ αξίες. Ο πολιτισμός και η ιστορία συνδέονται και θα πρέπει ο πολιτισμός ως αποτέλεσμα της ιστορίας να προστατεύεται. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες μέλη της, ε, μέλη της Ένωσης να βοηθήσουν τους νέους που συμμετέχουν στην πολιτιστική ε, βιομηχανία μέσω δράσεων στην παραγωγή, ε, στη διαχείριση και αλλού και βέβαια το Erasmus εδώ είναι μια καλή πρωτοβουλία που βοηθάει την πολιτιστική παραγωγή. Εγώ ίδια έζησα και σπούδασα και στις δύο υπήρες, υπήρους και κατάλαβα ακριβώς τη σημασία που έχουν οι πολιτισμικές ανταλλαγές και η κατανόηση, η αμοιβά κατανόηση των πολιτισμών. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας εταιρικής σχέσης Ένωσης Αφρικής θεωρώ ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές δεν θα πρέπει να είναι μονομερής και ότι η διάσπορα, η διασπορά συγγνώμη, θα πρέπει να μας επιτρέπει να έχουμε καλές, διά, καλούς διάβλους επικοινωνίας και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά. Θεωρώ λοιπόν ότι μέσω αυτής της δήλωση μπορούμε να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες για τους νέους και να αντιμετωπίσουμε πώς θέματα φύλου, αναπηρίας, γεωργικής ε, ε, συγγνώμη, καταγωγής. Αυτό που εμένα σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ και εγώ, λέει η πρόεδρος Κάμπερ Εβερτ. Ε, φτάνομαι στον τελευταίο ομιλητή τη σημερινή ε, ε, συνεδρίασης, ο κύριος Ματόκο, είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της UNESCO για την Αφρική. Έχει το λόγο αγαπητή κυρία. Ah, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω τα όσα ήδη λέχθηκαν. Νομίζω ότι υπάρχουν θεμελιώδη ερωτήματα που θέσανε οι ευρωβουλευτές σας και που χρειάζονται ίσως περισσότερη απάντηση είτε εδώ είτε αλλού και που θα πρέπει σε αυτά να βασίσουμε τον προβληματισμό μας για θέματα παιδείας και πολιτισμού. Ο πρόεδρος της ε, Νότιο Αφρικανικής Δημοκρατίας είπε χθε ότι η Αφρική ε, διαθέτει πολυφωνία και οι νεολαίες της το ίδιο και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρί νεότητα. Έχουμε την νεότητα τη υπαίθρου, των αστικών κέντρων, αυτή που έχει πέρασει από το σχολείο, αυτή που είναι προνομιούχα, αυτή που δεν είναι και βεβαίω και η διασπορά. Ανθρώπου νέου που ψάχνουν δουλειά και νέου και νέε που φτιάχνουν startup στην Αφρική. Όλη αυτή η νεότητα συνολικά έχει ανάγκη από στοχευμένες απαντήσεις. Έχουν και ένα κοινό ενδιαφέρον. Όλοι έχουν την ίδια επιθυμία. Θέλουν να χειραφετηθούν, θέλουν και πολιτικά να χειραφετηθούν, θέλουν να ε, χειραφετηθεί η Αφρικανική Ήπειρος, θέλουν να ε, υλοποιηθεί η Ατζέντα 2063, όπως είπε προηγουμένως η βουλευτής από την Ογκάντα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Ας υπενθυμίσουμε ορισμένους αριθμούς. Πρώτα, κάθε χρόνο 11 εκατομμύρια νέων μπαίνουν στην αγορά εργασίας και 4 εκατομμύρια είναι μεγάλη κατά μέσον όρο. Έχουμε ε, κάποια σχέδια για τους ανθρώπους αυτούς για να έλθω στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών. Τα εκπαιδευτικά μας συστήματα, η παιδεία μας ανταποκρίνεται, είναι προσαρμοσμένη ε, ε, στην απασχόληση που αναζητούν οι νέοι αυτοί. Υπενθυμίζω και την έκθεση του 1996 που πρόβλεπε τέσσερι σημαντικού πυλώνε. Γιατί και εμεί στην Αφρική του ξεχνούμε του πυλώνε αυτού. Η παιδεία δεν είναι μονάχα να μάθει κανεί να γράφει και να διαβάζει, αλλά να μάθει να γνωρίζει, να μάθει να κάνει πράγματα και να είναι συμμετοχή επομένω στη, στην κοινωνία και κυρίω να μάθει την συμβίωση. Απαντώ ε, έτσι σε αυτά που είπατε για τις συγκρούσεις ε, ε, ειρήνη κλπ οι απαντήσεις που δίνουμε είναι πάντοτε μερικού χαρακτήρα ή ανεπαρκής. Δεύτερο, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που ως UNESCO βλέπω ότι τα θέματα αυτά τονίζονται εδώ και κυρίως η εκπαίδευση των νέων κοριτσιών. 40% των νέων κοριτσιών που μπαίνουν στο σχολείο στις χώρες του Σαχέλ έχουν λάβει διεθνή στήριξη για την εκπαίδευσή τους. Ε, αλλά ε, δεν αρκεί αυτό. Ε, μιλήσαμε για ε, πολιτισμό, μιλήσαμε για αναγκαστικούς γάμους, μιλήσαμε για τον ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων που ξεπινούν από τον Τακάρ, ακόμα και από τα Αμπιτζάν. Σε 30 χιλιόμετρα μόλις φύγετε από τα αστικά κέντρα βλέπετε τα νεαρά κορίτσια που κουβαλάνε ε, ε, μεγάλους κάδους στην πλάτη για να πάνε να φέρουν νερό. Αυτά δεν γίνονται παντού, αλλά γίνονται σε πάρα πολλέ και σε μεγάλες πόλεις, στην Πραζαβίλη, στον Τακάρ για όσους γνωρίζουν τις περιοχές αυτές. Υπάρχουν σχολεία όπου τα νέα κορίτσια δεν μπορούν να πάνε σε τουαλέτες, σε αποχωρητήρια που να του προσφέρουν και κάποια προστασία. Μιλώ για τι κλασικές απαντήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εμεί, η UNESCO, και οι μη κρατικέ οργανώσει πρέπει να κάνουμε σημαντικέ εκστρατείε. Η παιδεία των κοριτσιών δεν είναι μονάχο αριθμό των σχολείων και των δασκάλων. Είναι μια πολιτιστική πρακτική που χρειάζεται, που μέχρι τώρα δεν επιτρέπει εύκολη πρόσβαση των κοριτσιών στην, ε, στην εκπαίδευση. Βουλευτή στο Νίγηρα που προσπαθεί να περάσει πρόταση νόμου στο κοινοβούλιο τη χώρα του για τους πρώιμους γάμους. Πέντε χρόνια παλεύει και παρά και τις πιέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν προχωρεί. Διότι όλοι 100% των βουλευτών εκεί είναι άνδρες και εμποδίζουν να προχωρήσει το σχέδιο νόμου. Οι γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια πρέπει να μπουν στα κοινοβουλευτικά σώματα. Πολύ σημαντικό. Είμαι επίσης ικανοποιημένο που είναι παρούσα η κυρία Κώστα την οποία είχα γνωρίσει όταν ήρθα εδώ την προηγούμενη φορά και μίλησε και για θέματα πολιτισμού και σε σχέση με την UNESCO. Έχουμε άλλωστε συμφωνίες συνεργασίας. Είναι σημαντικό διότι στην ε, συμφωνία, στην σύμβαση, ένας από τους τρόπους να προσεγγίσουμε την νεολαία είναι η ε, βιομηχανία πολιτιστικών. Έχετε το γνωστό ματονγκέ εδώ στις ε, Βρυξέλλες έχετε το 18ο ε, του Παρισιού. Οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπετε εκεί είναι καλλιτέχνε. Έτσι αυτό ορίζονται. Είτε πρόκειται για σχεδιαστές μόδας, είτε πρόκειται για τραγουδιστές, είτε πρόκειται για κομμωτέ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στην Ευρώπη για να βρουν απασχόληση στους τομείς αυτούς και τελικώς καταλήγουν να, μπουν, να γίνουν ή ε, θηροροί νύχτας. Ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, δημιουργικότητα αυτή και χρειάζονται και κοινοβουλευτικές δίωδοι και νομοθετικές δίωδοι που να επιτρέψουν την ενίσχυση του πολιτιστικού γίγνεσθε στην Αφρική. Χρειάζεται μια υποδομή πόσες, πόσα σχολεία καλλιτεχνών υπάρχουν στην Αφρική, πόσα σχολεία designer υπάρχουν στην Αφρική. Μαζί με τον κύριο Αλφαντή που είναι μεγάλος Αφρικανός σχεδιαστής και είναι και πρέσβης της UNESCO προχωρούμε στη δημιουργία μιας ε, σχολής μόδας στον Ιαμέη στην Αφρική. Πόσα σχολεία καλών τεχνών υπάρχουν στην Αφρική Θυμούμε τη σχολή του Πότο Πότο, στο Ντακάρ υπήρχε μια σχολή ε, ζωγραφικής. Είναι πολύ λίγες. Όλοι αυτοί οι νέοι ε, πάνε και φτιάχνουν ένα DVD, ένα CD ε, και τελικώ του εκμεταλλεύονται κιόλα. Χρειάζονται λοιπόν να δημιουργηθούν σχολέ, αλλά χρειάζεται και να του συνοδέψουμε από, από το Α μέχρι το Ω, από την αρχή τη καριέρα του μέχρι τη σύνταξή του. και οι λιγότερο νέοι Αφρικανοί που ε, είχαμε γνωρίσει την ε, σπουδαία αφρικανική μουσική γνωρίζαμε ότι οι καλλιτέχνες μας δεν είχαν απολύτως τίποτα και δεν έχουν και καμιά εξασφάλιση για τη μεγάλη ηλικία, ούτε στάξουν τίποτα. Δεν είναι νορμάλ πράγματα αυτά. Σήμερα υπολογίζεται 2-3% το ακαθάριστο προϊόν της ε, δημιουργικής βιομηχανίας. Δέστε τι γίνεται στις αφρικανικές πόλεις πόσοι άνθρωποι, πόσοι νέοι εκεί φτιάχνουν ε, μουσικά συγκροτήματα. Έχω πέντε ανήψια που πάνε σε σχολεία εμπορικά κλπ. Το μόνο που θέλουν όμως είναι να γίνουν ράπερ στο YouTube. Δεν έχουν τη στήριξη για να το κάνουν. Πέντε, πέντε ανήψια έχω. Ε, είναι πολλά, ε. Και κορίτσια μεταξύ τους. Πρόκειται για πράγματα που πρέπει να βάλουμε θεμέλια. Μη λησμονούμε και την νεότητα της διασποράς. Και όχι μόνο στην Ευρώπη βέβαια. Και σε ό,τι αφορά την συμμετοχή στα κοινά, εγώ λέω στους νέους, όλοι μας περάσαμε από την νεαρά ηλικία και όλοι διεκδικήσαμε τα δικαιώματά μας. Σεις που έχετε τώρα την τύχη να είστε μέσα σε ε, οργανώσεις, ούτε τα κοινοβούλια ούτε οι υπουργοί θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά στη ρίζα, στις τοπικές κοινότητες, στα χωριά. Ποιος δουλεύει για αυτούς, ποιος μεταφέρει τη φωνή τους. Δεν είναι οι νέοι που έχουν πρόσβαση στο YouTube και στο διαδίκτυο. Όλοι αυτοί οι νέοι, αλλά και οι νέε στα ε, κοριτσάκια που από τεσσάρων χρονών πάνε στα χωράφια να δουλέψουν, ε, να ε, συνοδέψουν τη μαμά τους στο πηγάδι του χωριού Ποιο θα απευθύνει το λόγο σε αυτά τα νέα παιδιά. Αυτό είναι μια δουλειά επίση που πρέπει να γίνει και να αναζητηθούν τα παιδιά αυτά και μέσα στι τοπικέ ε, ε, κοινότητες. Ο κ. Νε, ε, Νεκόφ είπε κάτι σχετικό. Εμείς για να πάμε σχολείο διανύαμε μια απόσταση 12 χιλιόμετρων. Τώρα όμως δεν χρειάζεται. Μπαίνετε στα, ε, ε, δίκτυα, στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπετε το Τόκιο χωρίς να χρειάζεται να πάτε ποτέ. για να μην μιλώ για UNESCO και για τον εαυτό μου το ίδιο, έχουμε ωστόσο δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο ενώσεων, οργανώσεων της νεότητας που δουλεύουν για την ειρήνη, για το ρόλο του πολιτισμού στην ειρήνη, κάνουν πολλές εκδηλώσεις και είναι και πολλές μάλιστα που εκπροσωπούνται και εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ελπίζω η συμβολή μου να κρυθεί θετική στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τους τρεις ομιλητές του δεύτερου γύρου έχουμε 21 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν είναι πολλά, αλλά θα προλάβουμε. Ο κύριος Βάκηλ ε, θα λάβει το λόγο. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας για την φτώχεια και την κοινωνική πρόνοια. Δύο λεπτά παρακαλώ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά κύριε Βάκη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συνάδελφοι ήδη μίλησαν για πολλά. Η εκπαίδευση στην Ιγυρία είναι υποχρεωτική και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έγιναν συντονισμένες προσπάθειες για σωστή παιδεία. Υπάρχει η Επιτροπή της Βασικής Εκπαίδευσης που ε, λαμβάνει υπόψη και θέματα ε, υποδομών για την παροχή της εκπαίδευσης. Έχουμε προβλήματα όπως αναφέρθηκαν. Έχουμε ανέργους νέους γιατί δεν έχουν δεξιότητες, δεν ξέρουν επαγγέλματα. Σε αυτούς τους τομείς μπορεί να παρέμβετε εσείς, να μας βοηθήσετε, ώστε η εκπαίδευση που θα δώσουμε στους νέους μας θα προσαρμόζεται προς τις επαγγελματικές ανάγκες, κυρίως τώρα στην παγκόσμια ψηφιακή εποχή. Στην Ιγυρία δημιουργούμε επίσης ε, και ε, εμπορικά κέντρα, ε, κέντρα εκπαίδευση, συγγνώμη, για να εξυπηρετηθούν οι νέοι. Στον αθλητισμό ε, μην ξεχνάμε νους υγιής εν σώματι υγιή. Πολύ σημαντικός ο αθλητισμός στην Ιγυρία και μας έκανε και ένδοξους με τους περίφημους αθλητές που αναδείχθηκαν σε πολλές αθλητικές κορυφές εκδηλώσεις. Πάρα πολλοί ε, ταλαντούχοι αθλητές είναι Νιγηριανοί και βεβαίως αυτοί προσδίδουν δόξα και στους νέους στη χώρα. Αυτό είναι κάτι που μας βοήθησε να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας ε, να δημιουργηθεί ένα κλίμα αδελφοσύνης ε, μεταξύ των νέων ε, και παροχή βοήθειας και συμπαράστασης. Εμείς έχουμε ε, σύνδεση με τις παραδόσεις μας. Σίγουρα όμως ε, θα πρέπει να αναζωογονήσουμε πολλές ε, από τις ικανότητες που διαθέτουμε. Με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Η Σαμπίνε Φερχάνη, δύο λεπτά. Καταρχήν ε, αυτό που διαπιστώσατε με λύπη ε, κυρία Φαμπρεγκέτ ότι δεν είμαστε πολλοί βουλευτές εδώ. Και εγώ λυπάμαι. Είναι πολύ κακό που δεν ε, αξιοποιούν όλες οι ομάδες την ευκαιρία αυτή. Οι μεγάλες ομάδες έχουν μια εκπροσώπηση, οι άλλοι όχι. Ε, και εγώ, ο συνάδελφος Νιζιντεύε, εγώ είμαι στην αντιπροσωπεία για την Νότια Αφρική και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Οπότε τουλάχιστον λίγοι είμαστε, αλλά είμαστε οι ειδικοί. Να πω κάτι. Όταν οι νεολαίστικες οργανώσεις κάνουν ε, πολιτικές δηλώσεις και περνούν ψηφίσματα, ε, αυτά λαμβάνονται υπόψη παρόλο που μπορεί να μην ε, αποτελέσουν αυτούσιες κομμάτι μιας νομοθετικής πρότασης. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε έχει την, το προνόμιο να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Αν εσείς δώσετε ψήφισμα στο Κοινοβούλιο, εμείς μπορούμε να το ε, συνεπεξεργαστούμε ε, παρόλο που δεν θα είναι αυτούσιο όπως είπα το νομοθετικό κείμενο και στο πλαίσιο της κανονικής νομοθεσίας κάποια θέματα ε, μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε. Είναι περίπλοκη διαδικασία και είναι δύσκολο και οι οργανώσεις νέων να παρακολουθήσουν μετά τι κάναμε μετά από αυτά που μας είπαν, αλλά μια καλύτερη επικοινωνία μπορεί να μας βοηθήσει να δείξουμε ότι αυτά που μας δίνεται δεν εξαφανίζονται, τα διαβάζουμε και όσο μπορούμε τα ε, ε, συμπεριλαμβάνουμε σε νέα νομοθετήματα για τον αθλητισμό θα ήθελα να ε, επανέλθω σε ένα θέμα. Όταν μιλάμε για αθλητισμό, ανάπτυξη και εκπαίδευση ε, ε, δεν σημαίνει ότι όλοι μέσα από αυτή την πολιτική θα, όλοι θα γίνουν επαγγελματίες αθλητές. Ο αθλητισμός όμως με την ευρεία έννοια είναι ένα βοήθημα για να μάθει κανείς και άλλα, άλλες δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, ακρίβεια, ε, φιλοδοξία. Υπάρχουν πολλά προγράμματα στην Αφρική που αποσκοπούν στην πρόληψη του AIDS και που περνούν μέσα από τον αθλητισμό. Έτσι περνάμε και κάποια στοιχεία κατανόησης ε, ε ορισμένων στοιχείων. Έτσι ο αθλητισμός λοιπόν μπορεί να ενταχθεί στην γενικότερη πολιτιστική πολιτική. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο να ε, ζητήσει κανείς ότι όλοι οι καλλιτέχνες από την Αφρική θα μπορούν να ε, εξασφαλίσουν ε, τον επιούσιο εδώ όλοι, αλλά καλό είναι να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, την ψηφιοποίηση ούτως ώστε να βελτιώσουν και στον πολιτιστικό τομέα την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους. Άλλωστε και εμείς στην Ευρώπη ε, ακολουθούμε παρόμοια συστήματα για να δώσουμε δυνατότητες στους δικούς μας καλλιτέχνες. Κυρία Κώστα, ευχαριστώ. Διάφοροι συνάδελφοι από εδώ ασχολούμαστε με το θέμα του πολιτισμού, της τέχνης και των γυναικών. Οπότε ελπίζω να είμαστε οι κατάλληλοι συνομιλητές για σας, αλλά και εγώ έλπιζα θα ερχόταν περισσότεροι συνάδελφοι. Χαιρετίζω και την κυρία Φαμπρικέτη, την οποία ήδη είχα συναντήσει σε ένα άλλο φόρουμ εδώ, και με συνάντηση στο Κοινοβούλιο και πραγματικά Εκτίμησα αυτά που είπε, όπως και αυτά που είπε και ο κύριος ο δόκτωρας Ματόκο. Τρία πράγματα να πω. Σήμερα νομίζω έχουμε καταλάβει, μετά από διάφορες τραγωδίες που συνέβησαν σε χώρες που μέχρι πρόσφατα ζούσαν πιο ήρεμα, ακλέφοντας του Κένια κτλ. Βλέπω λοιπόν ότι αν στο κέντρο ή στο επίκεντρο των πολιτικών της νέας εταιρικής ε, σχέσης είπε κτλ. Αν δεν βάλουμε λοιπόν στο επίκεντρο τον πολιτισμό, κινδυνεύουμε να χάσουμε άλλη μια γενιά νέων. Αν δεν αναγνωρίσουμε λοιπόν τον πλούτο που αντιπροσωπεύουν αυτές οι νέες γενιές. Και αυτό το 1,4 δις, είμαστε οι πρώτοι δωρητές, εντάξει, αλλά αυτό θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε πιο έντονα. Θα πρέπει επίσης να βρεθούν και μηχανισμοί, ενδεχομένως και κοινοβουλευτικοί, πέρα της ε, αντιπροσωπείας ΑΚΕ που έχουμε στο Κοινοβούλιο. Να δούμε πώς θα μπορούσαμε να παρενεύουμε μαζί με τις δηλώσει που κάνατε, ας πούμε, εσείς στη διασκέψη, στη διασκέψη κορυφής, ώστε αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική να πει στο επίκεντρο των προσπαθείο μας ε, παγκοσμίω ώστε να εμπλέξουμε και του τοπικού φορεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και από εσά μάλιστα, ώστε να δούμε ακριβώ ποιοι είναι οι πιο αξιόλογοι συνομιλητέ, ώστε να εμπλέξουμε και την κοινωνία των ε, πολιτών. Και νομίζω ότι πραγματικά εδώ έχουν στρατηγικό ρόλο οι νέοι τη διασπορά. Τέλο, η Αφρικανική Ένωση, οι διεθνεί οργανισμοί και αυτοί θα πρέπει να συμμετάσχουν πέραν του Κοινοβουλίου επειδή, όπως λέγαμε, η νομοθεσία για τις γυναίκες στην ε, Αφρική ή για την υποχρεωτική εκπαίδευση, τουλάχιστον στην ε, πρωτοβάθμια, θα πρέπει να επεκταθεί. Και εδώ ακριβώς θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσπάθεια διαφόρων διεθνών οργανισμών πάντοτε στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών της Αφρικής. Εμείς είμαστε πάντως διαθέσιμοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να δώσω ευχαριστώ πολύ να δώσω τον λόγο στον Τζόνσον Ουκούμα που είναι βουλευτής του ε, Κοινοβουλίου της Νιγηρίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εσείς οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές και άλλοι βουλευτές λέγομαι Ουγκούμα από την Νιγηρία. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμούμε με μεγάλη νοσταλγία όταν ήμουν μικρό παιδί είχα τόσους συγγενείς που είχαν πάει να σπουδάσουν στην Ευρώπη και στην Αμερική και στη Βουλγαρία και στη Ρωσία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τι έγινε εκείνη η πολύ ευγενική σας, ευγενή σας πολιτική που οδήγησε ε, σε τόσο σημαντικές προσωπικότητες που είχαν πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία σας. Δίνατε υποτροφίες και αυτές οι υποτροφίες έβγαλαν πολλούς από τη φτώχεια οι οποίοι μπόρεσαν να απολαύσουν μετά σημαντικότατη παιδεία. Θα πρέπει να κάνετε κάτι για να ενθαρρύνετε την αφρικανική νεολαία. Μην κλείνετε τις πόρτες σας απέναντι στους Αφρικανούς νέους. Αυτά που ακούτε για μετανάστευση Όλοι αυτοί θέλουν να έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά που έχετε δώσει στην Αφρική, για παράδειγμα, ως παιδιά. Για παράδειγμα, στο γυμνάσιο που πήγαινα εγώ, είχαμε υποστήριξη από την Αμερική και από αλλού. Και είχαμε, ε, για παράδειγμα, ε, ε, αθλητικό εξοπλισμό. Αυτά τα χρειαζόμαστε και τώρα και χρειαζόμαστε πρόσβαση και στην εκπαίδευση στην Αλοθαπή. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος Κάμερ Εύερτ. Θα παρακαλέσω τώρα να λάβει τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ την, την συναδελφό μου Κλέαρ Μορέλ που έδωσε πληροφορίες σχετικά με το τι κάνουμε ε, και τι κάνουμε και εμείς ως Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακή συνεργασία Μιλήσατε για την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία που αποτελεί και τον στόχο μας η ανάπτυξή της στη συνεργασία με την Αφρική. Μάλιστα σήμερα καθυστέρησα να προσέλθω εδώ διότι συζητούσαμε για μια χρηματοδότηση 15 εκατομμυρίων ένα πρόγραμμα που λέγεται επενδύσεις σε δημιουργικότητα και πολιτισμό και τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά κατευθύνονται σε νέους και νέες και ιδίως για identity building και sharing. Μια νέα προσέγγιση που προσπαθούμε να συνδέσουμε τις δεξιότητες που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο, πολιτιστικές, δημιουργικές κλπ, με την παγκόσμια αγορά και κοινωνία. Μία από τις αιτίες της μετανάστευσης δεν είναι μονάχα η έλλειψη απασχόλησης, αλλά και η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ίδια του τη χώρα και η έλλειψη ταυτότητας των ανθρώπων αυτών και η έλλειψη ας πούμε περηφάνειας για το πολιτιστικό τους υπόβαθρο. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να βασιστεί στις παραδοσιακές δεξιότητες και να συμβάλλει στη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας και αγοράς μιλούμε για identity building και sharing όπως είπα αυτή την κίνηση δηλαδή από την ύπεθρο στα αστικά κέντρα εκεί έχει και μια αρνητική πτυχή που είναι ότι χάνουν την πολιτιστική τους ταυτότητα και την διασύνδεσή τους με τις τοπικές κοινωνίες είπατε κι εσείς ότι ο πολιτισμός είναι το κατάλοιπο της ιστορίας Ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ε, συνεργαστούμε και με την UNESCO για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και το 2018 που θα είναι και έτος πολιτιστικής κληρονομιάς θα είναι και μια ευκαιρία, ένα πλαίσιο δηλαδή για να ε, αποδώσει η προσπάθειά μας. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα δύο παρεμβάσεις. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα λεπτό και πρώτη κυρία Σόιντροβα. Δεν είναι ερώτηση. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που δουλεύετε, συνεργάζεστε με τους ανθρώπους, με τον κόσμο τις χώρες σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έμφαση που δίνετε στους νέους και στην παιδεία. Νομίζω ότι στην ίδια κατεύθυνση κινούμεθα και εμείς επενδύσεις για τους νέους. Διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όπως είπατε εσείς από την Ιγυρία Ίσως χρειάζεται να επενδύσουμε περισσότερα στην υγεία, στα σχολεία, στα σχολικά κτίρια, στις αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ. Σας ευχαριστώ όλους και όλους. Και νομίζω ότι εμείς θα ε, ψάξουμε να επενδύσουμε στους νέους και στο μέλλον μας. Julie Ward, ένα λεπτό. Yeah, thank you for the... Ευχαριστώ πολύ για την συνέχιση της καλή συζήτηση και ο διαλόγο που έχουμε εδώ. Καταρχάς να πω πόσο καλό ήταν το η κυρία Williams της αναγνωρίστηκε η συμβολή και χαίρομαι γιατί είναι Βρετανή αφρικανικής καταγωγής. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για αυτήν. Χάρηκα που άκουσα την συζήτηση για τον αθλητισμό που όπως ξέρουμε έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι από την ε, εκλογική περιφέρεια του Μάτσεστερ και του Λίβερπουλ και όπου και να πάω λέω ότι είμαι από το Μάτσεστερ και όλοι με αναγνώριζαν αμέσω. Έχουμε βέβαια του γνωστού παίχτε, ακριβοπληρωμένου κλπ. Αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα αυτοί για να αντιμετωπίσουμε τι μορφέ ρατσισμού. Και θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση για το πόσο ευρύ είναι ο για τον αθλητισμό ή θα μπορούσε να είναι. Γιατί έχουμε πολλά, πολλές μορφές αθλητισμού, όχι μόνο ανταγωνιστικές. Να, να ρωτήσω και κάτι άλλο για την κυκλική οικονομία. Για τα θέματα του περιβάλλοντος που είναι πολύ σημαντικά για τους νέους. Τι γίνεται. Συγγνώμη που πρέπει να είμαι αυστηρή, δεν γίνεται αλλιώ. Έχουμε τέσσερα λεπτά για τρεις ομιλητές. Λοιπόν, πολύ σύντομα σε ένα λεπτό ή δυνατόν. Ξέρω ότι ζητάω το αδύνατον, αλλά τι να κάνουμε. Ποιος θα αρχίσει. Αρχίστε εσείς. Αυτός φοράει το καπέλο του και στο κρεβάτι για το θέμα της εκπαίδευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όντως, να αναπτύξουμε τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός πραγματικά βοηθάει τα παιδιά σε όλες τις χώρες. Without education, they are no redundant. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα επικεντρωθούμε κατά το ίμιση των αθλητισμών και το άλλο ίμιση στην εκπαίδευση για να προωθήσουμε ακριβώς όλες τις μορφές αθλητισμού σε επίπεδο συλλόγων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο αθλητισμός στην Ιγυρία θα είναι αποδεκτός από τον πληθυσμό. Αν το κάνουμε αυτό, ο κόσμος θα είναι απασχολημένος, θα απασχολείται αντί να κάθεται. Και αντιμετωπίζουμε και άλλα φαινόμενα εδώ, όπως ε, δραστηριότητε Μπόκο Χαράμ και τα λοιπά. Αυτά που με ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Α, ο κύριος Ματόκο. Ευχαριστώ, σύντομα. Για την νέα εταιρική σχέση που αναφέρθηκε. Είπε σε ένα πάνελ χθε ένα νέος Θερματολόγια άρα και δράση. Αλλά δράση από κοινού. Και η κυρία Μογκυρίνη είπε ότι πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αφρικανική Ένωση υπάρχουν και άλλοι διεθνεί οργανισμοί όπως ο ΙΕ που εργάζονται σε αυτό το πεδίο. Ας εργαστούμε λοιπόν από κοινού γιατί υπάρχουν όλα τα περιθώρια συνομιλίας και συνεργασίας υπέρ των νέων. Εγώ ως ε, πρόεδρος της να σας πω ότι είμαι... είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή τη δουλειά με όσο ενδιαφέρονται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Φαμπρικέτ, λέει πρόεδρος. Εκτός μικροφώνου, μικροφών τώρα, να ανακάνετε το ασύνηθες, να δώσω τον χρόνο μου στην Σίντια Μουκαντή, που είναι μια νέα επιχειρηματίας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, να σας δώσει δύο στοιχεία για τις ε, νέες αυτές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ όμως πάρα πολύ σύντομα. Ένα λεπτάκι έχετε. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Να μιλήσω γαλλικά. Βάλτε ακουστικά. Ναι, για τον πολιτισμό. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τα ψηφιακά θέματα, τα οποία είναι σημαντικά για την ανανέωση του πολιτισμού, επιτρέπουν τη διατήρηση του πολιτισμού, τη μετάδοση στην διασπορά, όπως επίσης και την ε, δημιουργία. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο κάτι το χειρονακτικό, αλλά και το ψηφιακό. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε τα θέματα τη εκπαίδευση στον πολιτισμό, γιατί υπάρχουν όλο και περισσότερε εφαρμογέ που πια σα επιτρέπουν να μάθετε να μετράτε, να διαβάζετε κτλ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τη διασπορά που μετά από την Ευρώπη θα τα μεταδώσει όλα αυτά στην Αφρική. Αυτά δηλαδή τα ψηφιακά μέσα. Θα μας βοηθήσουν όλα αυτά επίσης να εντάξουμε τις ε, γυναίκες, ώστε να γίνουν ένα πρότυπο για, τις, για τα μικρά κορίτσια, ώστε να τα βοηθήσουν να βρουν μια δουλειά στην Αφρική. Επίσης, σε επίπεδο εκπαίδευσης, μια και έχω πολύ χρόνο, να μιλήσω για την κινητικότητα και να πω ότι το το πρόβλημα για τις Αφρικανές είναι η θεώρηση. Αν έρθουν στην Ευρώπη θα πάνε αλλού. Ρωσία, Κίνα, Αμερική και αυτό θα μεγάλει πολύ άλλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και όλες σας. Για... Ευχαριστώ τους ομιλητές που μας ε, παρουσίασαν την κατάσταση στην Αφρική. Μας βοήθησαν πολύ. Να είστε βέβαιοι ότι και εμείς θα τα συμπεριλάβουμε αυτά στις περαιτέρω εργασίες μας παρόλο που μπορεί να μην γίνει ένα προς ένα και, όπως είπε και η συνάδελφος Σαμπίνε Φερχάιμ. Ε, σίγουρα οι αντικειμενικοί περιορισμοί καμιά φορά είναι τρομακτικοί, αλλά τι να κάνουμε υπάρχουν. Εμείς δίνουμε μάχες για περισσότερα κονδύλια και για την Ευρώπη και ε, δεν τα καταφέρνουμε πάντα όπως θέλουμε. Θέλω να μας πιστέψετε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όμως για να προχωρήσουμε εδώ. Ευχαριστώ θερμά και πάλι. Η επόμενη συνεδρίαση θα είναι σε 7 Δεκεμβρίου το απόγευμα από τις 3 μέχρι τις 6.30 το απόγευμα. Και ευχαριστώ θερμά και τους διερμηνείς μας που μας βοήθησαν πολύ. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Καλημέρα σε όλους.